προσωπίας που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Μας είπαν και αυτοί ότι θέλουν να αναβληθεί και ούτε και αυτοί μπορούν να είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να αναβληθεί η εξέταση της αναφοράς αυτής για τον Νοέμβριο, το σημείο 9 δηλαδή. Ε, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, λέει Πρόεδρος, προβλήματα γι' αυτό, αλλά βέβαια θέλω οι συνάδελφοι να πούν. Υπάρχει καμία αντίρρηση για την τροποποίηση αυτή στην ημερήσια διάταξη, να βγάλουμε το σημείο 9. Ωραία. Συνεπώς, κατά τα άλλα, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έρχομαι τώρα στο σημείο 2, που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 15 Ιουλίου 2010. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά, εφόσον δεν πείτε τίποτα στο μεταξύ στην γραμματεία. Ανακοινώσει του πρα... Ο κύριο Βίλαντ είναι σε αποστολή στην Αυστρία και ζητά συγγνώμη που δεν θα μπορέσει να είναι εδώ σήμερα. Μετά την ψηφοφορία πρέπει να ξέρετε ότι θα έχουμε μια σύντομη παρουσίαση από πλευράς του Αντιπρόεδρου Σεύκοβιτς. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λοιπόν, Μάρος Σεύκοβιτς, για πρώτη φορά μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ μαζί μας και να συνομιλήσουμε έτσι. Ξέρετε... Ότι... Γνωρίζετε ότι θέλουμε να υποβάλουμε ερωτήσεις αυτόν και ελπίζουμε ότι θα μας απαντήσει. Θα παραμείνει βέβαια για μαζί μας περίπου μία ώρα και έτσι θα ρυθμίσουμε και τον χρόνο παρέμβασής μας ώστε να μπορέσουμε από πλευράς επιτρόπου να λάβουμε απαντήσεις για, την πολιτική, για τον πολιτικό προσανατολισμό και επίσης ε, με μια συνομιλία με τα μέλη της Επιτροπής. Στον Επίτροπο επίσης την 10-28 2008 ε, για την ρύθμιση σε περίπτωση περιπτώσεις παραβίασης και την γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής, αυτήν αναφορά πάνω και όλα αυτά βρίσκονται στο φακέλου σας. Για να το δούμε λοιπόν αυτό το θέμα και μετά από τον Επίτροπο Σεύκοβιτς θα ξεκινήσουμε με τις συζητήσεις για τις αναφορές και θα είναι παρόντες ορισμένοι από εκείνους που έχουν υπογράψει αυτές τις αναφορές, κυρίως στο 10 την αναφορά επίσης το σημείο 11 και την αναφορά στο σημείο 12. Και για το σημείο 18 την γνωμοδότηση Άγκης για την ε, ελεύθερη πρόσβαση σε έγγραφα θα το μελετήσουμε αυτό και παρουσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Κάτι ακόμα να σας πω ότι πάνω σε αυτό το σημείο σημειώθηκε ιδιαίτερη εξέλιξη με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον Βαβάρια Λέγα και είχαν αλλάξει ορισμένα σημεία τα οποία ίσχυαν μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα εξετάσουμε και τις νέες αυτές εξελίξεις. Μετά από τη συνάντηση των συντονιστών ε, αύριο στις 5 θα ασχοληθούμε με την Ερευνητική Επιτροπή που είχε επισκεφθεί ήταν σε αποστολή και μετά θα έχουμε μια συνάντηση μαζί με την Επιτροπή ΑΦΚΟ και αυτό παρουσία των εκπροσώπων Εθνικών Κοινοβουλίων. Ακόμα θα έχουμε στο σημείο 21 στην ημερήσια διάταξη, την εξάρτηση του θέματος για το σύστημα εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακόμα κάτι, η 1665 στο σημείο 56 στο β σημείο αυτό δεν ισχύει πια. Ε, γιατί, γιατί έχουμε νέα στοιχεία από πλευράς υπογράφοντος την έκθεση αυτή. Και στο σημείο αυτό, αν δεν έχουμε άλλες ανακοινώσεις από πλευρά συναδέλφων, αν έχετε το λόγο. Στα διάφορα για αύριο, για την 1667 του 2007. Είναι μία αναφορά την οποία θα συζητήσουμε αύριο. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μπει σαν πρώτη στην επόμενη συνεδρίαση. Γνωρίζω πολύ καλά τα γεγονότα και στην περίπτωση αυτή πιστεύω ότι πρόκειται για αποζημίωση εξόδων και τα λοιπά. Θα ήθελα λοιπόν και αυτό να μπει σαν α, στην κατηγορία των αναφορών α. Εντάξει, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο γιατί μου υπενθύμησε έτσι αυτό που θα πρέπει να παραλαμβάνω κάθε τόσο για τις αναφορές που έχουν εγγραφεί στο Β το παράρτημα ότι θα ε, αντιμετωπιστούν έτσι με τον τρόπο αυτό αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από πλευρά συναδέλφων. Γι' αυτό να έρθουμε τώρα στο σημείο 5 θα ψηφίσουμε την ε, ετήσια έκθεση Μάλλον θα εξετάσουμε την, της έκθεση του Ευρωπαίου Διασυλλομιβητή για το έτος 2009, Ντεντέλσεβα, η συγγήτρια και αν δεν θα ήθελα να πει κάτι η συγγήτρια, να περάσουμε στην ψηφοφορία και μάλιστα αμέσω. Ναι, μπορούμε, μπορούμε. Ξεκινάμε αμέσως με την ψηφοφορία. Μία και μόνη τροπολογία. έχει να κάνει με την παραγραφό 16. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία αυτή. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την έκθεση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με μία αποχή. Ψηφίζουμε την πρόταση αυτή μετά την τροποποίησή της. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται μία και μόνο αποχή. να ευχαριστήσω την συνάδελφο Δεντέλτσεβα για την εργασία της και να έρθουμε τώρα στο σημείο 6. Είναι η έκθεση επί της ειδικής εκθέσης που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβήτης κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγγελία 676 του 2008 η κυρία Παλιαδέλη είναι η συγγήτρια. Θα ήθελα να τη ρωτήσω, θα ήθελα να πει κάτι σχετικά. Uh, Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής για την βοήθειά τους, τη συνεισφορά τους. Και αυτή η έκθεση που δεν τροποποιείται, ίσως μπορεί να θεωρηθεί σαν έγκριση της όλης ιδέας. Γεγονός είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε το έργο του διαμεσολαβητή και ελπίζω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να το δείξουμε αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω κατάλογο ψηφοφοριών. Έχετε εσείς κάποιο κατάλογο ψηφοφοριών. Εγώ δεν έχω. Είναι πρώτη φορά που θα ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι. Οπότε δεν ξέρω τι κάνουμε καμία τροπολογία, γι' αυτό ψηφίζουμε μόνο το ψήφισμα ως έχει προταθεί. Η σκιώδη συγγήτρια κυρία Μπαζέσκου. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι όπως γνωρίζετε δεν έχουμε τροπολογίες και αφού δεν έχουμε τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης το ΕΛΚ υπερψηφίζει, εγκρίνει δηλαδή. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την έκθεση αυτή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Μία αποχή. Ευχαριστούμε την συνάδελφο Μπαλιαδέλη και την κυρία Μπαζέσκου. Το σημείο 7 τώρα, γνωμοδότηση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι η συγγήτρια με μία τροπολογία από πού ξεκινάει αυτό, από πού προέρχεται μάλλον από μια συμβιβαστική λύση για τη δική μου τροπολογία και συναδελφού Μάγερ ψηφίζουμε ψηφίζουμε παρακαλώ τη συμβαστική αυτή λύση, πρόταση παράγραφος 4 υπέρ παρακαλώ κατά τις αποχές σας Εγκρίνεται. Μία αποχή μόνο. Ψηφίζουμε την γνωμοδότηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση αυτή με μία αποχή. Και να που τελειώσαμε με το θέμα των ψηφοφοριών. Τώρα ακρόαση με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς που μας είχε πει ότι θα έλθει εδώ στις τρεις και μισή. να όμως που εμείς είμαστε πιο γρήγοροι και από τη σκιά μας και έτσι δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, συγγνώμη μια στιγμή. Από ό,τι με ενημερώνουν, ίσως έλθει λίγο νωρίτερα ο Επίτροπος, ε, γι' αυτό λιγόλεπτη διακοπή περιμένοντας τον Επίτροπο. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Μάρο ε, που είναι εδώ μαζί μας ε, και το χαρτοφυλάκιο του είναι οι θεσμικές ε, σχέσεις και η διοίκηση. Θα ήθελα να αναγνωρίσω και να συγχαρώ τον κύριο Σεύκοβιτς ε, γιατί ιδιαίτερα ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στις σχέσεις με την Επιτροπή μας και μάλιστα πριν από τον ορισμό του σαν Επιτρόπου και ε, ερχόταν σε επαφές ε, με την Επιτροπή μας που μερικές φορές ε, δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη από την Εκκληστική Επιτροπή. Και τον Ιούλιο που μας πέρασε ήλθα σε επαφή με τον Επίτροπο, συναντήθηκα μαζί του και του έθεσα ορισμένα θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας και μας απασχόλησαν αρκετές φορές όπως το κύριο θέμα που είναι μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην δική μας την Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάναμε από κοινού μια εκτίμηση της καταστάσεως και ότι απαιτείται ένας διάβλος επικοινωνίας και να μπορέσουμε έτσι να είναι και πιο χρήσιμη και λειτουργική η επικοινωνία αυτή που και τα όσα λέμε εδώ να περνάν και παρά έξω. Αυτά λοιπόν θα έχει τον λόγο επίτροπος, μετά θα του υποβάλλετε ερωτήσεις και μετά θα απαντήσει εκείνος. Ο Επίτροπος έχει το λόγο και τον ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία του εδώ ανάμεσά μας. Thank you very much, uh, Madam Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την πρόσκλησή σας. Έχω προσπαθήσει να ακολουθήσω τις παραδόσεις του προηγούμενου επιτρόπου και επίδειξα φορά φράγματα για να καταφέρω να φτάσω εδώ παρόλο που είναι κλειστή η δρόμη και είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς ε, εδώ από την Επιτροπή. Τα κατάφερα όμως και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Με βοήθησε εδώ και η συνάδελφος. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να μιλήσω μαζί σας για θέματα που αφορούν τους πολίτες και να συζητήσουμε μαζί και άλλα ζητήματα. Πήρα κάποιες ερωτήσεις από εσά που έχουν να κάνουν κυρίως με την πρωτοβουλία πολιτών. Θα σας μιλήσω λοιπόν γι' αυτό, θα σας πω που βρισκόμαστε, ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο και επίση θα σα πω ότι προσβλέπω συνεργασία με τη δικιά σα την Επιτροπή ώστε να προχωρήσουμε και να ολοκληρωθεί η συζήτηση για το θέμα αυτό της πρωτοβουλία Ευρωπαίων ε, πολιτών και να γίνει μια πραγματικότητα. Την Άνοιξη είχα πάρα πολύ δουλειά με την πρωτοβουλία αυτή. Βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέστηκε πολύ από την Ισπανική Προεδρία να προχωρήσει ε, με τις προετοιμασίες για την πρόταση αυτή κανονισμού. Είχαμε μια έντονη συζήτηση επίσης με το Συμβούλιο που κατέληξε σε μια γενική πολιτική συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε είχε πει ότι πρέπει να πάρουμε το χρόνο μας, ότι πρέπει να έχουμε έναν πολύ καλό κανονισμό για να βοηθήσουμε τους πολίτες να επικοινωνούν καλύτερα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ξέρετε ότι ορίστηκαν το καλοκαίρι οι εισηγητές και είχαμε έναν άτυπο τριμερή διάλογο την προηγούμενη εβδομάδα μόλις. Πού βρισκόμαστε λοιπόν τώρα. Πρέπει να σας πω ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους προχωράμε. Όπως γνωρίζετε, η συνθήκη είναι αρκετά λακωνική όταν μιλάει για την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Μιλάει, λέει ότι πρέπει να είναι ένα σημαντικό αριθμό πολιτών από διάφορες χώρες μέλη. Εμείς τώρα πρέπει να αποφασίσουμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό, τι σημαίνει ε, μεγάλος αριθμός ε, πολιτών, ε, χωρών, τι σημαίνει αυτό. Είπαμε κάποια στιγμή για ένα εκατομμύριο υπογραφές. Έτσι λοιπόν τώρα ερχόμαστε στον αριθμό των χωρών μελών πόσες πρέπει να είναι. Λέμε ότι πρέπει να είναι το 1 τρίτο. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι το 1 τρίτο γιατί αυτό φαίνεται λίγο στην ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας γιατί το ίδιο ισχύει για να δημιουργηθούν ομάδες για την ενισχυμένη συνεργασία. Για παράδειγμα επίσης χρειάζεται το 1 τρίτο των χωρών μελών για να έχουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς επικουρικότητας κτλ. Δηλαδή σε διάφορους τομείς το βρίσκουμε αυτό το 1 τρίτο στη συνθήκη. Για μας όμως, όταν μιλάμε για το 1 τρίτο των ε, χωρών, το λέμε γιατί θέλουμε αυτή η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών να είναι πραγματικά Ευρωπαία. Δεν θέλουμε να πρόκειται για μια περιφερειακή πρωτοβουλία, τοπική πρωτοβουλία που να ενδιαφέρει λίγου μόνο σε μια γωνιά τη Ευρώπη. Όχι, θέλουμε το 1 τρίτο των χωρών. Πιστεύουμε τότε είναι πραγματικά ευρωπαϊκό το αίτημα. Και γιατί. Γιατί με την πρωτοβουλία αυτή θα οδηγηθούμε ενδεχομένω σε νομοθεσία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις 27 χώρες μέλες. Οπότε πρέπει να είναι πολύ καλό να έχουμε μια στέρεα βάση με μεγάλη υποστήριξη από το 1 τρίτο των χωρών μελών. Και επίτα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ξέρετε και εσείς δηλαδή καλά, ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση είναι πολύ δύσκολο και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το εξή. 0,2% του πληθυσμού μιας χώρας φτάνει, δεν είναι αρκετό. Αν έχουμε πάρα πολλές ε, υπογραφές από την Γερμανία και πολύ λιγότερες από μικρές χώρες, το Λουξεμβούργο για παράδειγμα, ε, χίλιες υπογραφές μπορεί να είναι αρκετές, αλλά έτσι δημιουργείται μια κατάσταση όπου ε, αν μιλούσαμε για νούμερα δηλαδή, οι μικρές χώρες θευνούνται σε σχέση με τις μεγάλες. Γι' αυτό προτιμούσαμε το ποσοστό. Έπειτα πολλαπλασιάσαμε τον αριθμό των ευρωβουλευτών και φτάσαμε στα νούμερα τα οποία σταθμίζουν κάπως τη διαφορά ανάμεσα σε μικρές ε, και μεγάλες χώρες. 72.000 για τη Γερμανία και 4.000 για το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα βάση του υπολογισμού αυτού με το 1 τρίτο. Για την ηλικία τώρα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε τη συμμετοχή των νέων. Να συμμετέχουν οι νέοι στη διαδικασία αυτή. Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο στην Αυστρία ψηφίζουν οι νέοι από τα 16. Στις υπόλοιπες χώρες μέλη ψηφίζουν από τα 18. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο μια χώρα να επαληθεύσει τις υπογραφές ατόμων οι οποίοι δεν είναι ακόμα ψηφοφόροι, δεν έχουν φτάσει στην ηλικία να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Έρχομαι τώρα και στον μηχανισμό της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Τα έχετε ακούσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ευρωβουλευτές αλλά και από τους πολίτες ότι θέλουμε έναν μηχανισμό που να είναι φιλικός προς τον πολίτη, εύκολος για τους πολίτες. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν του πώς θα ε, συμπεριλάβουμε τους πολίτες, πώς θα παληθεύσουμε τις υπογραφές τους κτλ. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να ξεκινήσει από τη στιγμή που περνάει στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, Γιατί τότε υπάρχει διαφάνεια, διότι εμείς ζητάμε κάποια ελάχιστα δεδομένα για να συμπεριληφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, το στόχο, το όνομα των οργανωτών και επίσης ποια είναι η χρηματοδότησή τους. Γιατί και αυτό χρειάζεται για να υπάρχει διαφάνεια. Πρέπει να ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί την πρωτοβουλία. Όταν έχουν γίνει όλα αυτά, τότε οι οργανωτές μπορούν να αρχίσουν με τη συλλογή υπογραφών. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σχεδιάζοντας ε, τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό, πώς αυτός να είναι εύκολος για τον πολίτη, φιλικός, αλλά και πώς να περιορίσουμε τις καταχρήσει. Να μην δημιουργήσουμε δηλαδή μια πλατφόρμα μέσα από την οποία οι οργανωτές να μπορούν να προχωρούν σε αντιευρωπαϊκές επιθέσεις ή να χρησιμοποιούν την πρωτοβουλία αυτή σε βάρος ευρωπαϊκών αξιών. Ή από την άλλη θέλουμε να δούμε πώς θα αποφύγουμε η πλατφόρμα αυτή να χρησιμοποιηθεί για να κορυδεύει κάποιος τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε πρωτοβουλίε οι οποίες πάνε σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια άλλη συζήτηση που κάναμε που ήταν πολύ δύσκολη ήταν για το αποδεκτό. Πότε είναι παραδεκτή και πότε όχι μια πρωτοβουλία. Υπήρξαν διάφορες σχολές σκέψεις. Ορισμένοι θέλαν να υπάρχει αυτός ο έλεγχος του παραδεκτού ήδη από την αρχή, πριν αρχίσει η συλλογή υπογραφών. Εμείς είπαμε ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή που θα οδηγήσει στη λήψη κάποια απόφασης, με περίπλοκα μάλιστα ζητήματα πολλές φορές, όταν δεν είμαστε προηγουμένως σίγουροι για την σοβαρότητα της πρωτοβουλίας και του οργανωτή. Να μην θέλουν δηλαδή να υποβάλουν αίτηση για μια τέτοια πρωτοβουλία απλώ και μόνο για να κάνουν διαφήμιση για του αυτού του ή για να κερδίσουν κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό θέλαμε να γίνεται έλεγχος από την αρχή και ότι από τις 180.000 τελικά υπογραφές αποφασίσαμε να αρχίζει αυτός ο έλεγχος. Ενώ στην αρχή η ιδέα ήταν για πάνω από 300.000 υπογραφές. Κάτι άλλο τώρα για την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε είναι να συζητήσουμε πώς ε, κρίνονται οι αιτήσει που γίνονται και οι οποίες τελικά δεν είναι παραδεκτές. Ποια θα είναι τα κριτήρια. Είπαμε όταν είναι αντιευρωπαϊκές, όταν είναι εκτός αρμοδιοτήτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα άλλο σωρό κριτήρια τα, αποφασίσαμε. Ελπίζω ότι θα, θα καταλάβετε όλα αυτά και θα στηρίξετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά εμείς θα θεωρούμε διοικητική απόφαση σε εκείνο το στάδιο. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, το μηχανισμό αυτών στο τέλος. Γιατί θα έχουμε χάσει πολύ χρόνο και πολλές προσπάθειες. Οπότε πρώτα παίρνουμε τη διοικητική αυτή απόφαση την οποία, με την οποία κανείς μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να προσφύγει αν θεωρήσει ότι δεν είναι σωστή. Πάντως προσπαθούμε εμείς να βρούμε και τρόπους να βοηθήσουμε τους οργανωτές κάθε φορά που θέλουν να συμπεριλάβουν μία πρωτοβουλία. Να τους πούμε τι πληροφορίες χρειάζονται, να τους συμβολέψουμε για την αρμοδιότητα. Όταν λοιπόν έχουν γίνει αυτά, τα κράτη-μέλη αρχίζουν να παληθεύουν ε, τις υπογραφές και υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Πάντως τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για το πώς θα παληθεύσουν τις υπογραφές. Δεν μιλάμε για δημοψήφισμα, δεν μιλάμε για εκλογές, οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και ε, σε στατιστικό επίπεδο, σε τυχαίο επίπεδο την επαλήθευση των υπογραφών. Αλλά αυτό θα το αποφασίζουν τα κράτη-μέλη κάθε φορά. Πόσε υπογραφές θα επαληθεύουν και με ποιο τρόπο. Έπειτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τέσσερι μήνες για να ε, εκδώσει μια ανακοίνωση. Η πρωτοβουλία πολιτών σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν τέτοια δικαιώματα όπως τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία αποφασίζουν για τους νόμους. Η Επιτροπή από τη δικιά της την πλευρά με το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχει αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Πάντως, σας διαβεβαιώ ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι αν έχετε μια πρωτοβουλία ενός εκατομμυρίου πολιτών που έρχονται από τα ένα τρίτο των χωρών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει κάποιο μήνυμα έτσι κι αλλιώ ήδη με αυτό. Οπότε θα φροντίσει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει έχοντας συνείδηση ότι υπάρχει πίεση από τον κόσμο να δουλέψει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Συγχρόνως οι πολίτες και εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται. Άρα η αντίδρασή μας θα είναι μία ανακοίνωση με την οποία θα σας εξηγούμε σε εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο κοινό πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοβουλία αυτή που έχει καταχωρηθεί. Την τελευταία φορά, κυρία Πρόεδρε, συζητήσαμε μαζί για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ρόλο της δικιάς σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην όλη διαδικασία. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εξαιτία της φύσης της δουλειάς σας εξαιτίας της φύσης των καθημερινών σας δραστηριοτήτων που είναι να λαμβάνετε αναφορές και να τις επεξεργάζεστε, βρίσκουμε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, άπαξ και έχει συμπληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης μιας ε, ε, πρωτοβουλίας και υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εις το μεταξύ. Φυσικό λοιπόν βρίσκω εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να οργανώνεται κάποια δημόσια κρόαση με τους οργανωτές της εκάστοτε πρωτοβουλίας, όπου να συζητιούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην πρωτοβουλία και ποιες είναι οι προσδοκίες των οργανωτών και των πολιτών. Έτσι, αν μη τι άλλο το κοινό θα αντιλαμβάνεται τις προσπάθειες που εμείς κάνουμε και που είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε, εφόσον έχουν κινητοποιηθεί τόσοι πολλοί πολίτες υπέρ της ε, όποιας πρωτοβουλίας. Θέλουμε λοιπόν να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσα από τη δικιά σας ε, επιτροπή να κινητοποιηθεί ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των οργανωτών για κάθε πρωτοβουλία. Δύο τελευταία σημεία που θέλω να θίξω, για τα οποία ξέρω ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, η συλλογή online. Και το δεύτερο είναι η προστασία των δεδομένων. Για τη συλλογή online πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στην συλλογή υπογραφών. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και την τεχνολογία στη πρωτοβουλία αυτή των πολιτών. θέλουμε να συμπεριλάβουμε τους νέους. Όταν λοιπόν έχει συμπεριληφθεί η online συλλογή, τότε βέβαια το ζήτημα τίθεται τι σύστημα θα χρησιμοποιήσετε και πώς θα προστατεύσετε τα δεδομένα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να ετοιμάσει ένα open source software που θα φοδώνουν οι οργανωτές για τη συλλογή των υπογραφών. Αυτό το software, αυτό το πρόγραμμα, θα καταχωρείτε και θα πιστοποιείτε για να ε, συλλέγει τα στοιχεία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον τομέα αυτό. Προστασία των δεδομένων αυτή καθεαυτή, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτες δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Υπάρχουν άρθρα που έχουν ετοιμαστεί σε συνεργασία με ε, τις υπεύθυνε αρχές για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φροντίσουμε λοιπόν τα κείμενα που θα υιοθετηθούν να συναδούν πλήρως με τα κείμενα που ήδη ισχύουν στο τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φροντίσουμε και για το θέμα της ευθύνης, πάντα σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει και θα προβλέψουμε και διαδικασίες ε, δίωξης εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα τα δεδομένα, εφόσον γίνεται καταχρησή τους, κάποιος τα πουλάει, κάποιος τα χρησιμοποιεί. Εδώ χρειαζόμαστε ένα πολύ στέρεο σύστημα διαφύλαξη δεδομένων, γιατί όταν μιλάμε για ένα εκατομμύριο υπογραφές, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τι κάνουμε με τα δεδομένα αυτά. Ελπίζω λοιπόν η αρχική πρόταση να αποτελεί όντως ένα πολύ καλό σημείο κίνησης. Καταλήξαμε εκεί αφού συζητήσαμε με το Συμβούλιο. Τώρα συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους εισηγητές σας πάνω σε αυτό και πολύ σύντομα θα έχουμε και τον επίσημο τριμερή διάλογο με την Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τις σωστές απαντήσεις στις απορίες μας και στα προβλήματά μας και να εγκριθεί το θέμα αυτό τον Δεκέμβριο στην Ολομέλεια, ώστε οι πολίτες να έχουν στη διαθεσή τους ένα νέο μηχανισμό επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω ότι μακρηγόρησε ήδη αρκετά. Είμαι στη διάθεσή σας για απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας δώσατε χρησιμότατες πληροφορίες και μας ανακουφίσατε με ορισμένα μας είπατε έτσι αρκετά νωρίς. Συνάδελφος, έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ επικοδομητική ατμόσφαιρα και κλίμα συζητήσεων αυτής της πρώτης ε, συνάντησης με την παρουσία της Βελγικής Προεδρίας και των ε, εισηγητών. Πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό ιονός για τις μελλοντικές μας ε, συναντήσεις αλλά και για την εμπιστοσύνη που θέλουμε να διοχετεύσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχει ένα έτοιμο κείμενο. Οι συνάδελφοί σαφώς θα γνωρίζουν ότι αυτή είναι η φιλοδοξία της Επιτροπής μας να διασφαλίσουμε ένα εργαλείο το οποίο θα είναι φιλικό προς τον χρήστη, προς τον πολίτη της Ευρώπης. Όλα αυτά τα χρόνια η Επιτροπή μας λαμβάνει αναφορές από τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι ένα διαφορετικό δικαίωμα το που έχουμε, το οποίο όμως ε, μοιάζει με αυτό που συζητάμε σήμερα. Εδώ αναφερόμαστε σε όλους τους ε, διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς απολύτως κανένα όριο ηλικίας και το δικαίωμα να ε, υποβάλουν αναφορές. Εδώ βεβαίως πρόκειται για μια δημόσια συζήτηση και το όριο ηλικίας στο 16ο όριο ηλικίας είναι κάτι που βεβαίως μπορεί να μας προβληματίσει. Από τη μία μπορούμε να πούμε ότι μη Εάν ε, μειώσουμε το όριο ηλικίας, ε, μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει Λέγοντα ότι οι νέοι, νέοι στην Ευρώπη, ε, όλο και νωρίτερα εμπλέκονται σε αυτήν την συζήτηση και τη δημόσια ζωή και ότι ενδεχομένω κινητοποιούμε το ενδιαφέρον. Δηλαδή δίνουμε δυνατότητες σε άτομα να υπογράψουν, να υποβάλουν στο όνομά τους μία αναφορά. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν πρέπει να γίνει διάκριση εδώ μεταξύ του ορίου ηλικίας το οποίο δίνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες για να ψηφίσουν και το όριο για να υποβάλουν και να υπογράψουν μία αναφορά. Το θέμα της πρώτης φάσης της καταχώρησης μιας αναφοράς. Συμφωνώ μαζί σας ότι εδώ ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας πρώτης επαλήθευσης, ενός πρώτου ελέγχου διοικητικού και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να το προτείνει και να δεσμευτεί η Επιτροπή. Το θέμα της επαλήθευσης των υπογραφών με συντομία. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Διότι από τη μία λέμε ότι είναι αρμοδιότητα κρατών μελών, ναι, το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα όπως ξέρετε κάποιων κρατών μελών που μπορεί να ζητήσουν ε, αποδεικτικά στοιχεία, ε, απόδειξη της ταυτότητας κτλ. Πράγμα το οποίο θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τη δυνατότητα υπογραφής μιας αναφοράς. Και το ερώτημα, που δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, είναι γιατί να περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Γιατί να ζητούμε στοιχεία ταυτότητας, παραδείγματο χάρη. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι βεβαίως η απέτηση αυτή μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό στοιχείο για κάποιον ο οποίος αρχικά επιθυμούσε να υπογράψει μία αναφορά. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά. Τι ακριβώς απαιτούμε από κάποιον ο οποίος θέλει να υπογράψει μία αναφορά. Και αντιθέτως να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να υπογράψουν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πολλά κρατημέλη και το δικό μου βεβαίως, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν πρόκειται να ζητήσει τέτοια χαρτιά ταυτότητας. Από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά και απαιτήσει και προϋποθέσεις που ισχύουν, δεν θα είναι ευρωπαϊκό εγχείρημα η υποβολή μιας αναφοράς. Το θέμα της δημόσιας ακρόασης. Ναι, βεβαίως όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το οργανώσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Αναφορών. Σαφώς και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε μια δημόσια κρίση. Οι περισσότεροι όμως από εμάς θεωρούν ότι εσείς η Επιτροπή είστε αυτοί στους οποίους απευθύνονται καταρχήν αυτές οι αναφορές. Και γι' αυτό και η αντίδραση και η απάντηση θα πρέπει καταρχήν να προέρχονται από εσάς. Η Επιτροπή λοιπόν ενδεχομένως θα είναι αυτή που θα πρέπει να σκεφτεί την δυνατότητα οργάνωσης μιας τέτοιας δημόσια κρόσης, από τη στιγμή βεβαίως που η πρωτοβουλία ε, συγκεντρώσει το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Εσείς είστε αν θέλετε ο κύριος ε, αποδέκτης, αυτόν στον οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο η αναφορά. Και βεβαίω αυτό μπορεί να γίνει μόνο και εφόσον εξετάσουμε προηγουμένω το περιεχόμενο μια αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πέτροπε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, αλλά να σας πω ότι είσαστε αποτελεσματικός, έγκαιρα ετοιμάσατε την πρωτοβουλία αυτή και να ξέρετε ότι όλοι μας υποστηρίζουμε τις προτάσεις σας, προτάσεις που ανταποκρίνονται απόλυτα στις δικές μας επιθυμίες. Μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατόν πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό η δικιά μας Επιτροπή να έχει λόγο σε αυτό το διάστημα κατά το οποίο εμείς μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούμε να ετοιμάσουμε την απάντηση, το σχέδιο απάντησης τέλο πάντων που προτείνουμε σαν λύση στο πρόβλημα που θα έχει θίξει η εκάστοτε πρωτοβουλία των πολιτών. Ευχαριστούμε. Γκόμς, η συνάδελφος. Thank you very much. Ε, ε, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε και δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και χαίρομαι γιατί ακούω ότι λαμβάνετε υπόψη σας θέματα που είχαμε υποβάλει, όπως παραδείγματο χάρη η μείωση των απαραίτητων ε, υπογραφών που μειώνονται από 500.000 εγώ άκουσα όμως και κάποιες άλλες προτάσεις για να είναι παραδεκτή μια αναφορά που χαμηλώνουν ακόμα περισσότερο το κατώτατο όριο. Επίσης το θέμα του ορίου ηλικίας. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται, πρέπει να είναι το ίδιο με το, την ηλικία των 18 ετών που ψηφίζουν οι νέοι πολίτες. Το θέμα επίσης της πρωτοβουλίας. Να βάλουμε λοιπόν όριο ηλικία, να μην βάλουμε. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Ξέρετε όμως ότι και το όριο ηλικία για τις εκλογές δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες. Θα ήθελα επίσης να σας υποβάλω και μία ιδέα η προστασία των δεδομένων, η ασφάλεια των δεδομένων για τους πολίτες της Ευρώπης είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε εδώ κάποια ασφάλεια όσον αφορά δηλαδή την καταχώρηση των αναφορών και όσον αφορά τις ε, τα στοιχεία που δίνουν οι πολίτε. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει ο θεματοφύλακα να είναι η Επιτροπή. Εκείνη θα δίνει εγγύησει όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία αυτών των προσωπικών δεδομένων. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία. Μπορούμε σαφώ ε, να συμφωνήσουμε μαζί σα όταν λέτε θέλετε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδου και να δημιουργήσουμε κάτι που να είναι πολύ πιο φιλικό προς τον χρήστη. Τι όμως εννοούμε φιλικό προς τον χρήστη. Νομίζω ότι έχουμε ιδέες εδώ στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει προηγουμένως να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Thank you. Mr. Commissioner... Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το πώς κρίνεται το σοβαρό μιας πρωτοβουλίας. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι αντικειμενικός ο κριτής ή η διαδικασία που θα κρίνει κατά πόσο μία πρωτοβουλία που προτείνεται είναι σοβαρή ή όχι. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Γιατί για τους Ευρωπαίους πολίτες η αντικειμενικότητα είναι κάτι πολύ βασικό. Κατά την περίοδο καταχώρησης μιας πρωτοβουλίας είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια που θα αποφασίσουν αν μια πρωτοβουλία είναι σοβαρή ή όχι. Η συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπο, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί είστε εδώ μαζί μας σήμερα και επίσης για όλες αυτές τις ιδιαίτερα λεπτομερείς πληροφορίες που μας δώσατε για το θέμα αυτό, για αυτή την πρωτοβουλία και να, τις διάφορες φάσεις συμφωνούμε όλοι μας ότι αυτή η πρωτοβουλία για τους πολίτες είναι μια σημαντικότατη διάσταση δημοκρατική στα δημοκρατικά μας όργανα και για τους πολίτες που θέλουν να δουν να εφαρμόζουν εφαρμόζεται αμέσως αυτή η πρωτοβουλία και να είναι απλή, σαφής, διάφανη η όλη διαδικασία. Να σας δώσω ε, συγχαρτήρια για τα όσα ακούσατε, ακούσαμε από εσά για τις αξίες μας, ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι στα αρμόδια της Επιτροπής και σε ευχαριστώ για τους συναδέλφους που online υπέγραψαν, υπογράφουν και ότι έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες πολιτών και ακόμα τρία θέματα, τρεις ερωτήσεις για τις τρεις φάσεις για αυτή την πρωτοβουλία για τους πολίτες, για τη φάση πρώτα απ' όλα για την καταχώρηση, για την αποδοχή και μιλήσατε για μια διοικητικής φύσεως επίσημη απόφαση από πλευρά Επιτροπής και τώρα τα κύρια αντεπιχειρήματα είναι ότι είναι και κριτής ε, και διαιτητής. Ε, τι κάνει η Επιτροπή ακριβώς ε, για να ανταποκριθεί, για να απαντήσει αυτό, τι γίνεται μια Επιτροπή Σοφών, μήπως για να αποφύγει αυτές τις κριτικές που καταλαβαίνουμε κατά κάποιο τρόπο πού οφείλεται αυτή η κριτική. Δεύτερο ερώτημα τώρα για τη φάση συλλογή και επαλήθευσης των υπογραφών, το εξέτασαν οι συνάδελφοι, γιατί έχει να κάνει βέβαια και με την προστασία των δεδομένων. Τι κάνει η Επιτροπή ίσως ένα περισσότερο δεσμευτικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων παρομοίων ε, και παρά το ότι η συλλογή και ο έλεγχος των υπογραφών θα γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Τι εννοούμε εθνικό επίπεδο διαφορετικό σε κάθε χώρα από τις άλλες. Ε, τι έγινε, ε, όπως το είχε προτείνει η Επιτροπή για ορισμένους περιορισμούς, τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε εσείς αυτό το άρθρο πώς ακριβώς έχει και για τη ρήτρα ευθύνη των κρατών. Σίγουρα χαιρόμαστε και ευχαριστούμε την Επιτροπή που το έχει συμπεριλάβει στο όλο θέμα. Και ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με την τελευταία φάση. Από τη στιγμή που θα περατωθεί η διαδικασία, τι θα γίνει, υπάρχουν δυνατότητες συγκεκριμένε ενδεχόμενα πλευράς Επιτροπής για να δούμε τις δύο δυνατότητες εάν ε, αυτή τη έχουν συλλεχθεί αυτές οι, επιτροπές, οι υπογραφές και αν δεν έχουν συμπληρωθεί. Τι θα γίνει, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να οργανώσει ακροάσεις και επιτρέψτε μου, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόμοιο μέσο και εργαλείο, ο ρόλος της Επιτροπής αναφορών πιο συγκεκριμένα, ποιος θα είναι στο ξεκίνημα, στην κατάληξη όλες διαδικασίες και για τις ακρόώσει, αυτά τα public hearings είναι ακόμα μια διαδικασία που ακολουθεί συνήθως η Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ. Ε, Ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, αλλά κάτι που δεν έχει να κάνει με την πρωτοβουλία των πολιτών. Κύριε Επίτροπε, εποφελούμε εδώ από την παρουσία σας ε, για να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα που εξετάσαμε εδώ. Είναι το προσωπικό με συμβασιούχοι εδώ στην Ευρωπαϊκή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίθετα με άλλους εργαζόμενους, αυτοί οι συμβασιούχοι έχουν σύμφωνα με τον κανονισμό τα ίδια δικαιώματα όπως και οι μόνιμοι υπάλληλοι, αλλά μπορούν να συμμετέχουν και σε εσωτερικούς διαγωνισμούς. Αυτό όμως είναι ε, κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σεβόμαστε έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο τέλος του 2012 θα ξεκινήσουν θεωρητικές εργασίες του κανονισμού αυτού. Πριν ξεκινήσουν από πλευράς Επιτροπής Ευρωπαϊκής αυτές οι εργασίες, θα πρέπει να κάνετε κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια, κυρίως για το άρθρο 9 του κανονισμού υπαλλήλων. Οι εσωτερικοί διαγωνισμοί εδώ, ε, εκεί έχουν πρόσβαση μόνο οι ε, όσοι έχουν προσωρινή συμβόλαια ε, και η μόνιμοι πάλι, όχι όμως έτσι συμβασιοχή. Ε, Και τώρα είναι περίπου το 20% του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως ε, και έτσι υπάρχει μία, ασκείται μία πολιτική διάκριση και επίσης χάνονται χρήματα για την πρόσληψη αυτή και υπάρχουν και πολλοί καταπιεσμένοι που υποφέρουν, που τους βλέπουν ότι απλά τους θεωρούν ξεχωριστά απ' έξω κανένα ξένο σώμα. Με την αλλαγή αυτή, την αναθεώρηση του άρθρου, θα μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν έτσι σε αυτές τις εσωτερικές διαδικασίες και διαγωνισμούς και διαφορετικά δεν θα πρέπει να ισχύει πια αυτός ο θεσμός του εσωτερικού διαγωνισμού. Να μας πει ο Επίτροπος τη φρονή σχετικά. Θα επανέλθω πάλι στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Εκπροσωπώ τους πρασίνους και έχω κάποιες ερωτήσεις. Έχετε βοηθήσει πολύ σε όλη τη διαδικασία και σας ευχαριστούμε. Το εκτιμάμε όλος ιδιαίτερο. Αλλά ας δούμε τα δύο επιχειρήματα. Μιλάτε για το 1 τρίτο των χωρών. Και αντιλαμβάνομαι το επιχείρημά σας, τη λογική του ότι πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία, να είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ναι. Αλλά τότε περιορίζουμε πάρα πολύ τις δυνατότητες. Για έξι χώρες είναι πολύ δύσκολο να μπουν μαζί Δέκα χώρες, που είναι το 1 τρίτο, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Υπάρχουν τόσο πολύ διαφορετικές νοτροπίες, ε, συνήθειες. Εδώ, με την πρωτοβουλία αυτή, πρέπει να μπορούν να έχουν μια φωνή άνθρωποι. Γιατί το δυσκολεύεται τόσο πολύ. Μόνο κάτι οι οργανώσεις όπως είναι εκείνες προστασίες των ζώων, ας πούμε, θα μπορούν να υποβάλουν πρωτοβουλίες που να κρίνονται παραδεκτές. Δεν είναι σωστό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται απαγορευτική πρωτοβουλία για πάρα πολύ κόσμο. Και σε σχέση με αυτό, κατάλαβα το επιχείρημά σα για το τρίτο, παρόλο που όπω σας είπα πιστεύω ότι είναι δύσκολο. 16 χρονών εδώ δεν ψηφίζουν, δεν πρόκειται για δικαίωμα ψήφου. Είναι για να αποφασίσουν κάτι και να αποφασίσουν κάτι θεωρούμε ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν κάτι και δεν θέλουμε να δεχτούμε το 16. Μα εμείς θέλουμε, τους ζητάμε να συμμετέχουν. Και έτσι κι αλλιώ μέχρι να προχωρήσει η περισσότερη πρωτοβουλία θα έχουν κλείσει όλοι τα 18, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Θα έχουν περάσει δύο χρόνια. Αν λοιπόν εσείς μπορούσατε να μου υποσχεθείτε ότι δεν θα έχουν κλείσει τα 18, καλά, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχουν φτάσει τα 18. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας επίσης ότι το κοινοβούλιο είναι τόσο δημοφιλές. Και παντού σε όλες μας τις χώρες χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα το δημοκρατικό αυτό θεσμό υπέρ της Ευρώπης. Λέμε ότι είμαστε δημοκρατικοί. Θα ήταν μια πολύ ωραία χειρονομία προς τους νέους αν τους λέγαμε «Ελάτε, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε». Και δεν πρόκειται για ψηφοφορία. Οπότε για ξανασκεφτείτε το. Μήπως τελικά μπορέσετε να πείσετε και την Επιτροπή να έρθει πιο κοντά σε μας. Δεν είσαστε και το πιο αγαπημένο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο στους νέους σήμερα, οπότε για κάντε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν θα έχω να κάνω με την πρωτοβουλία πολιτών τα ερωτήματά μου να σας ρωτήσω μερικά πράγματα για, για το Costa στην Ισπανία, Παράλληλα γιατί εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαστε με αυτό, είναι ευαίσθητο το θέμα και έχει να κάνει και με το δικαίωμα ιδιοκτησίας γενικά στην Ευρώπη. Η Επιτροπή Αναφορών ε, ζήτησε την νομική άποψη της νομικής υπηρεσίας ε, για το συμπεριληφθείς ε, στην συνθήκη της Λισαβόνα ε, το θέμα αυτό σχετικά με τη διακτησία, αλλά τι γίνεται, ήδη διατύπωσε μια γνωμοδότηση η Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό. Κάτι ακόμα, ένα δεύτερο ερώτημα για την πρόσβαση στα έγγραφα. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εργάζονται σχετικά με αυτό τον κανονισμό για την πρόσβαση και στην Μπαβάρια λέγεται η Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδίκα στην απόφαση ε, σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δικαιωμάτων ε, στοιχείων. Εδώ ξέρετε κάτι σχετικά και ακόμα από πλευράς Επιτροπής Ευρωπαϊκής ίσως υπάρχει ένας κοινό δρόμος για να μπορέσετε να ενημερώνετε τους πολίτες ε, γιατί το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ε, σχετικά με τον Μεσολαβητή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι ακριβώ γίνεται σχετικά. Ναι, συνάδελφε, έχετε το λόγο. Yes, before I start, ε, Πριν ε, ξεκινήσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Επίτροπε, και εσάς και όλους τους συνεργάτες σας για την εξαιρετική το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας ε, που δείξατε. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε και να μάθουμε πολύ από αυτό. Βασιζόμαστε στην υπάρχουσα κατάσταση και θα πρέπει από εδώ και πέρα, βασιζόμενοι στην υπάρχουσα εμπειρία, να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο το οποίο θα οδηγήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική. Η συνάδελφος έκανε ένα πολύ ε, ενδιαφέρον ερώτημα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς τα έξω. Θέλουμε να καλέσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ή θέλουμε να τους εμποδίσουμε από το να ε, χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Και εδώ θα αναφερθώ σε κάποιους κανονισμούς. Καταρχήν, όλα όσα αφορούν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις Επιτροπής, θέματα δηλαδή για τα οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορούν θέματα πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Μήπως όμως θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση νωρίτερα και να μην περιμένει 300.000 ή 200.000 υπογραφές γιατί από ό,τι φαίνεται θα πρέπει πρώτα να κινητοποιηθούν 100, 200, 300 άνθρωποι και μετά να πούμε σταματήστε, πρώτα θα ελέγξουμε το κατά πόσο αυτή η αναφορά είναι παραδεκτή, αν μπορεί να γίνει δεκτή και κατόπιν μπορεί ενδεχομένως να πούμε ότι η διατύπωση δεν είναι υπρέπουσα, ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί κτλ. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε πολύ νωρίτερο στάδιο ήδη από την αρχή και βέβαια να μην επιτρέπουμε σε κάποιο οργισμένο Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίο κάτι άκουσε στην τηλεόραση παραδείγματο χάρη και χωρίς να γνωρίζει ακριβώς περί τίνο πρόκειται, να ξεκινάει με μια τέτοια πρωτοβουλία. Η πρότασή μου είναι να υπάρχει ένα είδο οργανωτικής επιτροπής που να συμπεριλαμβάνει μέλη από διαφορετικά κράτη-μέλη. Τα άτομα δηλαδή να πρέπει να συναντηθούν, να σκεφτούν λίγο όρημα το τι θέλουν να υποβάλουν, να σκεφτούν τη διατύπωση και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως θα γινόταν και ένα ξεκαθάρισμα για το τι θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αλλιώ τους σταματάμε κάπω στη μέση και ο έλεγχος γίνεται σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο. Και αυτό νομίζω δεν είναι ε, ικανοποιητική διαδικασία. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, και εδώ ξέρω ότι οι παραδόσεις διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ξέρω ότι σε πολλά κράτη-μέλη όμως θα δημιουργήσουμε πρόβλημα εάν όποιος υπογράφει καλείται να υποβάλει και τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει μεγάλη αντίθεση. Υπάρχουν χώρες στις οποίες ε, ψηφίζουν οι άνθρωποι στα δημοψηφίσματα χωρίς να υποβάλουν κανένα αποδεκτικό ταυτότητας. Και πιστεύω ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα προτιμήσουν να μην υπογράψουν μία αναφορά παρά να υποβάλλουν ε, τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Το θέμα λοιπόν της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και ο αρμόδιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων ε, είχε ακριβώς αυτή την θέση, ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, είναι σαν να ζητάμε ποιος ακριβώς υποστήριξε μια συγκεκριμένη αναφορά. Δεν μας αφορά αυτό. Εμείς αυτό που θα πρέπει να ελέγξουμε είναι πόσοι, πόσους Ευρωπαίους πολίτες αφορά. Και κάτι άλλο που έφυξε και κάποιος άλλος συνάδελφος είναι το θέμα του χρόνου. η χρονική περίοδος που θα ορίσουμε, κατά την άποψή μου και σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε, νομίζω ότι ένας χρόνος είναι αρκετή χρονική περίοδος για ένα κράτος μέλος. Για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πιστεύω ότι είναι πολύ λίγο. Και δεν θα φτάσουμε σε αυτές τις 180.000 υπογραφές γιατί θα περάσει το 12 μήνο και δεν θα έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των υπογραφών. Πιστεύω ότι θα πρέπει λοιπόν, όπως ξέρετε υπάρχει διαφορετική διαδικασία αν πρόκειται για υπογραφές online είτε στο χαρτί. Πάντως για υπογραφές στο χαρτί ο ένας χρόνος δεν αρκεί. Και ένα άλλο ερώτημα είναι τελικά γι' αυτό το ένα εκατομμύριο υπογραφές που θα συγκεντρωθούν σε κάποιες περιπτώσεις, τι θα είναι το αποτέλεσμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δέσμευση, κανονισμός, ε, τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. πιστεύω ότι θα πρέπει να οδηγήσει μια τέτοια πρωτοβουλία που συγκεντρώνει ένα εκατομμύριο υπογραφές σε μια συζήτηση, σε ένα διάλογο. Μια διαδικασία αποδεκτή και από τους μεν και από τους δε και εν πάση περιπτώσει μήπως αυτό θα ήταν και μια εξαιρετική ευκαιρία για σας, για την Επιτροπή έτσι ώστε να εκφράσετε τις απόψεις σας, τις ιδέες σας στο κοινό. Αν λοιπόν ε, όντως ένα θέμα συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές, δεν θα ήταν η ευκαιρία να καλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Πιστεύω ότι με αυτού του είδους την συνεργασία θα δημιουργήσουμε όντως ένα κείμενο, ένα κανονισμό, ο οποίος θα είναι ευανάγνωστος και φιλιππικός προς τον πολίτη. να λάβει το λόγο ο Επίτροπος για να απαντήσει, να ρωτήσω κάτι σχετικά με τις διαδικασίες επί ε, λάβαμε μια αναφορά που ζητάει μια αναθεώρηση του μηχανισμού για παραβάσεις ε, που δείχνει ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα μπερδεμένα και δεν επιδιώκουν πραγματικά τους στόχους που θα θέλαμε να πετύχουμε και για παρόμοιο θέμα, για παραβάσεις είχαμε αρκετές φορές σαν Επιτροπή Αναφορών ζητήσει μια σχετική συνεργασία με την Επιτροπή Ειδικότερα όταν για τις διαδικασίες για παραβάση εκεί έχουν να κάνουν και αναφορές που μπαίνουν στη μέση και αυτό για να μην γίνει μάται η εργασία μας. Έτσι εσείς τι φρονείτε σχετικά. Ευχαριστούμε και έχετε το λόγο κύριε πίτροπε. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους όσοι πήρατε μέρος στη συζήτηση. Υπογραμμίσατε τα σημαντικά για σας, αλλά σημαντικά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σίγουρα και για το Συμβούλιο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τελικά είναι την καλύτερη δυνατό λύση για την πρωτοβουλία των πολιτών. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα για την κυρία Wallis. Συνεργαζόμαστε σε πολλά θέματα μαζί κυρία Wallis και εγώ. Οπότε καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία σας και καταλαβαίνω και γιατί κι άλλοι επιμένουν τόσο πολύ ώστε η πρωτοβουλία των πολιτών να γίνει όσο γίνεται πιο πολύ ελκυστική για τους νέους και όσο γίνεται πιο εύχρηστη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό λοιπόν και προσπαθούμε να πετύχουμε τα 16 χρόνια σαν όριο ηλικίας αποδεκτό για την υπογραφή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Πρώτα απ' όλα ακούσαμε τα κράτη-μέλη, τα οποία θέλουν να επαληθεύουν τις υπογραφές. Και από αυτά που μας είπαν καταλάβαμε, και σίγουρα και στην τριμερή συζήτηση θα το ξαναπούνε, Καταλάβαμε λοιπόν ότι για αυτούς τα κράτη-μέλη είναι δύσκολο να επαληθεύουν αν τα άτομα που θέλουν να επαληθεύσουν δεν έχουν κλείσει τα 18, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου δηλαδή. Λένε ότι τους είναι πολύ δύσκολη η, η επαλήθευση συγγνώμη, των υπογραφών σε αυτή την περίπτωση. Και σίγουρα υπήρξε και ενα πολιτικοφιλοσοφικό θέμα που συζητήθηκε. Έχουν δικαίωμα να είναι πολιτικά δραστήριοι οι νέοι άπαξ και δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν. Προσπαθώ να σας εξηγήσω πώς καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θα το θέσετε και πάλι και θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε στον τριμερή διάλογο το θέμα του ορίου ηλικίας. Σύντομα. Το ίδιο ισχύει και για την επαλήθευση διαβατήριο, ταυτότητα. Στην Επιτροπή πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το περίπλοκο παράρτημα ε, στο οποίο καταλήξαμε μετά από την Γενική Συμφωνία με το Συμβούλιο. Και αυτό γιατί κάνει την πρωτοβουλία Ευρωπαίων ε, πολιτών να φορτώνεται με διάφορα παράρτηματα, ε, με διάφορες περιπτώσεις στην κάθε χώρα. Βέβαια η κάθε χώρα προσπαθούσε να συμπεριλάβει πώς θα μπορούσε καλύτερα να επαληθεύσει. Άλλα θέλει η Εστονία που μίλησε για κάτι δικά διαβατήρια που έχουν ναυτική, άλλοι για τις ταυτότητες. Φτάσαμε στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι αρχές θέλουν μέσω των τοπικών αρχών και των δήμων που κατοικούν οι υπογράφοντες να μπορούν να παληθεύσουν τις υπογραφές. Προσπαθήσαμε έπειτα να βρούμε μια λύση για όλα αυτά, ζητώντα την άποψη των εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη. Τι δεδομένα χρησιμοποιούν συνήθω για να επαληθεύουν τι υπογραφέ. Και στο τέλο καταλήξαμε με το παράρτημα που περιλαμβάνει τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αλλά συμφωνώ ότι καλό θα ήταν να το ξαναδούμε. Συμφωνώ επίσης με την κυρία Wallis για το ότι σε μας απευθύνονται οι πολίτες με την πρωτοβουλία τους αυτή. Άρα εμείς πρέπει να απαντάμε και στους ε, οργανωτές της εκάστοτε πρωτοβουλία. Θα το κάνουμε, δίχως άλλο. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο κύριος Σέφνερ σε μια ακρόαση, εδώ καλό θα ήταν να μπορέσουμε και εμείς να παρουσιάσουμε την ανακοίνωση που θέλουμε να έχουμε, την διαδικασία που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Έχουμε κάποια εμπειρία για το πώς να προετοιμάσουμε τον κανονισμό αυτό. Κάθε φορά που ετοιμάζουμε μια νομοθεσία, στρεφόμαστε στους ενδιαφερόμενους στα διάφορα μέρη που θα κληθούν να εφαρμόσουν την κάθε νομοθεσία άπαξ αρχίσει να ισχύει και ξέρουμε ότι υπάρχει μια ποικιλομορφία θέσεων, ιδέων και απαντήσεων κάθε φορά που προτείνεται μια νομοθεσία. Οπότε εννοείται ότι και θα ερχόμαστε σε επαφή με τους οργανωτές. Αν έρθει για το περιβάλλον, για παράδειγμα, μια ε, πρωτοβουλία πολιτών και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο τομέας από τον οποίο θα έχουμε τις περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι φυσικό να ζητήσουμε από τους οργανωτές και από τα διαφερόμενα μέρη να έρθουν και να συζητήσουμε μαζί πριν να καταλήξει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να υπάρχει μια τέτοια επαφή δηλαδή πριν. Θα συνεχίσω τώρα με τον Βίκτορ Μπουστινάρο. Ευχαριστώ πολύ για την στήριξη. Συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας, άπαξ και εγκριθεί ο κανονισμός για την πρωτοβουλία πολιτών και θα ξέρουμε πώς η συνεργασία αυτή θα μπορεί να προχωρήσει συγκεκριμένα. Η κυρία Γκένς τώρα αναφέρθηκε στο παραδεκτό της πρωτοβουλίας. Αναφέρθηκε σε ένα software open source. Πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε με την έννοια αυτή του παραδεκτού. Και είναι κάτι που το ζήτησε και το Κοινοβούλιο και ε, συζητήθηκε στις διαβουλεύσεις που είχαμε με τον κόσμο. Οπότε, Εμείς αυτό που θέλαμε είναι να ξέρουμε ότι οι οργανωτές δεν μαζεύουν εις μάτι τις υπογραφές. Θέλουν να ξέρουν ότι θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, άρα ότι νομικά στέκει. Συζητήθηκε κατά πόσο θα πρέπει να γίνεται ο πλήρης έλεγχος στο αρχικό στάδιο ή όχι είπαμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια κατάχρηση. Γιατί μπορεί να προσπαθήσει κάποιος να καταχωρήσει μια πρωτοβουλία και να ξεκινήσουν συζητήσεις χωρίς να είναι σίγουροι οι οργανωτές ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τον αριθμό των υπογραφών ή ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία έτσι κι αλλιώς για άλλους λόγους. Προχωράμε με την ιδέα που σας πρότεινα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι πρέπει να ξεχάσουμε λιγάκι το παραδεκτό ή όχι, τον έλεγχο δηλαδή αυτόν, να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο στάδιο της καταχώρησης και μετά να δούμε το παραδεκτό ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι κοιτάμε να μην είναι κατά των ευρωπαϊκών αξιών ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η πρωτοβουλία. Επίσης ότι η πρωτοβουλία ε, δεν είναι δεν ε, κατέχεται από έλλειψη σοβαρότητας. Και το τρίτο κριτήριο που νομίζω ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν καταχωρούμε πρωτοβουλίες που είναι εκτός αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή πρωτοβουλίες για τις οποίες έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορέσει να προτείνει νομοθετική ρύθμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν χρειάζονται αυτά τα τρία κριτήρια, να γίνονται αυτοί οι τρεις έλεγχοι. Άπαξ και έχουν γίνει, τότε οι οργανωτές μπορούν να είναι περίπου σίγουροι ότι άπαξ και έχουν συλλέξει τις υπογραφές και έχουν υποβάλει την πρωτοβουλία αυτή, η πρωτοβουλία θα είναι παραδεκτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα την επεξεργαστεί και θα φροντίσει να νομοθετήσει σύμφωνα με την επιθυμία των οργανωτών. Θέλουμε να διευκολύνουμε λοιπόν τους οργανωτές, αλλά θέλουμε να διευκολύνουμε και τη δικιά μας τη ζωή της Επιτροπής. Γι' αυτό και μιλάμε για διοικητική απόφαση, δηλαδή οι υπηρεσίε θα εγκρίνουν τη διαδικασία, δεν θα περνάει από όλη τη διαδικασία για να φτάσει στο σώμα των επιτρόπων. Και ότι απόφαση έτσι κι αλλιώς πάρει η Επιτροπή, αν θέλει κάποιος μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Υπάρχει δηλαδή εγγύηση για τους οργανωτές ότι δεν θα είναι μόνο η Επιτροπή που θα αποφασίζει για το παραδεκτό ή όχι, είναι κάτι που μπορεί να το προσβάλλει κανείς στο δικαστήριο. Κύριε και τώρα ρώτησε για την σοβαρότητα, η τιμή σοβαρότητα μιας πρωτοβουλίας. Frivolous στα αγγλικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα μου ότι κάποιος ε, θέλει να προτείνει έναν ροκστάρ για πρόεδρο της Επιτροπής ή κάτι άλλο που δεν είναι καθόλου σοβαρό. Αυτό φαίνεται από την αρχή. Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο αυτό για να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις πρωτοβουλίες, απλώς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε να τηρήσουμε τα κριτήρια που έχουμε βάλει. Και είπαμε ότι αν δεν συμφωνούν οι οργανωτέ μπορούν πάντα να προσφύγουν στο δικαστήριο και να πούνε ότι α, εδώ η Επιτροπή δεν τηρεί σωστά τα κριτήρια. Αλλά τέτοιου παραμέτρου θέλουμε να του χρησιμοποιούμε γιατί αλλιώ ποιο ξέρει τι πρωτοβουλίε θα μας φτάσουν που δεν θα είναι καθόλου σοβαρές. Δεν θα ήταν καλό κάτι τέτοιο. Για το software open source. Εδώ έχουμε ακούσει πολύ προσεκτικά τα σχόλια των Ευρωβουλευτών και των κρατών μελών ότι για τους οργανωτές είναι πολύ πιο εύκολο να κατεβάζουν ε, open source software και έτσι να μπορούν να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα για κάθε πρωτοβουλία πολιτών. Οπότε έτσι η διαδικασία προχωράει πολύ πιο γρήγορα και είναι πιο εύκολο και η Επιτροπή να επεξεργάζεται την όλη διαδικασία μέσω ενός τέτοιου προγράμματος. Η κυρία Ντότζοβα τώρα. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. για την συλλογή online. Όπως είπα, καταλήξαμε ε, σε αυτό γιατί θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία. Όπως επίσης, επειδή προχωράει πιο γρήγορα και πιο εύκολα η διαδικασία όταν γίνεται συλλογή υπογραφών online. Και προσελκύει και περισσότερο τους νέους. Είναι πιο ελκυστική μια τέτοια online συλλογή υπογραφών για τους νέους. Ξέρετε πόσο χρόνο τρώνε στα Twitter και στα Facebook και σε άλλα ε, κοινωνικά δίκτυα οι νέοι. Οπότε πολύ πιο εύκολα θα χρησιμοποιήσουν μια τέτοια πλατφόρμα ξέροντας ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορη διαδικασία από ότι αν γραπτά πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους. Τώρα, για την άλλη ιδέα που ακούστηκε, ότι η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει αν είναι παραδεκτή, καταχωρήσιμη, για να το πω αλλιώς, μια πρωτοβουλία. Αν είμαστε μόνο εμείς που θα μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο, καταλαβαίνετε ότι έτσι μπορεί να καθυστερήσει πολύ διαδικασία. Καταλαβαίνω λοιπόν την ιδέα αυτή για μια επιτροπή σοφών που λέτε, αλλά η Γενική Γραμματεία μας να ξέρετε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους οργανωτές να προετοιμάζουν, να διατυπώνουν και να καταχωρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Βρίσκω ότι αυτό είναι καλύτερη ιδέα από το να προσθέσουμε ένα νέο σώμα που θα εξετάζει το παραδεκτό ή το καταχωρήσιμο μιας πρωτοβουλίας πολιτών. Για το θέμα της ρήτρα ευθύνη δεν έχω το κείμενο μαζί μου, αλλά αυτό που λέει το άρθρο είναι ότι κάθε οργανωτής είναι υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία στη χώρα που συλλέγουν τις υπογραφές. Είναι αστική ευθύνη αλλού, αλλού είναι πρόκειται δικήματα, αν δεν υπάρχει προστασία των δεδομένων τα κράτη-μέλη έχουν τη δικιά τους νομοθεσία για να αποφασίσουν τι γίνεται αν υπάρξει παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Κάποια φορά είπα ότι στον κανονισμό θα υπάρχει υποχρέωση η Επιτροπή να ρωτάει τους οργανωτές πώς θέλετε να συνεχίσετε. Να υπάρχει επαφή για να υπάρχει καλύτερη κατανόηση. Τρία σενάρια βλέπω εγώ. Να προχωρήσουμε όπως θέλουν οι οργανωτές να προχωρήσουμε, με νομοθετική πρόταση. Μπορούμε όμως και να το αρνηθούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πρωτοβουλία μπορεί να είναι παραδεκτή, μπορεί να ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά να μην θέλει να δώσει συνέχεια η Επιτροπή. Το παράδειγμα που δίνω είναι την κατάργηση της ε, άδεια Ορισμένοι μπορεί να μην τη θέλουν. Και τι θα γίνει λοιπόν. Άρα πρέπει να έχουμε την ευχαίρεια να αποφασίζουμε αν θα δώσουμε συνέχεια ή δεν θα δώσουμε συνέχεια σε μια τέτοια πρωτοβουλία πολιτών. Ή μπορεί να αποφασίσουμε για κάποιες τροποποίησεις ή να πούμε ότι θέλουμε επιπλέον πληροφορίες πριν δώσουμε συνέχεια στην πρόταση της πρωτοβουλίας. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες, ένα φάσμα δηλαδή ε, δυνατοτήτων που έχουμε για να δώσουμε συνέχεια στην πρωτοβουλία. Ένα εκατομμύριο υπογραφές από πολλές χώρες μέλη δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι μεγάλη πίεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προφανώς και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή για να δει τι τη ζητάνε οι πολίτες και άρα τι θα κάνει. Για τους συμβασιούχους. Η ερώτηση του κ. Βαλέσα. Γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εσωτερικούς διαγωνισμούς οι συμβασιούχοι. Εδώ η κατάσταση έχει ως εξής. Οι εσωτερικοί διαγωνισμοί, και εδώ σας τα λέω από μνήμης, θα σας το δώσω και γραπτά αν θέλετε, πάντως το βασικό είναι ότι οι εσωτερικοί διαγωνισμοί είναι για τους υπαλλήλου, για τους μονίμους υπαλλήλου, για τους υπολλήλους που έχουν περάσει διαγωνισμό και έχουν προσληφθεί οι οποίοι έχουν την πιστοποίηση ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να είναι μόνιμοι υπάλληλοι και μετά πάνε στους εσωτερικούς διαγωνισμούς. Οι συμβασιούχοι δεν περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Και δουλεύουν και σε διαφορετικές θέσεις συνήθως. Για τους συμβασιούχους ισχύει ότι ένας από τους επικεφαλείς είναι μόνιμος υπάλληλος. Είναι διαφορετική δηλαδή η διαδικασία από την οποία περνάει ο συμβασιούχο και ο μόνο υπάλληλο. Γι' αυτό και δεν μπορούν οι συμβασιούχοι να συμμετέχουν στου εσωτερικού διαγωνισμού που προβλέπονται για του μόνιμου. Αλλά θα συζητηθεί το θέμα του κανονισμού για το προσωπικό. Γιατί το 2012 λύγει και η συμφωνία για του μισθού. Ξέρω ότι θα γίνουν και γίνονται ενδιαφέρουσε συζητήσει και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τι δημοσιονομικέ πρόπτικες. Οπότε θα ακουστούν πολλά ενδιαφέροντα εκεί. Θα το ξαναδούμε δηλαδή. Θα δούμε τον κανονισμό προσωπικού. Και πάλι. Ο οποίο πρέπει να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι κι άλλιω. Το κάνουμε αυτό για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Αλλά μέχρι να υπάρξει τροποποίηση, ό,τι ισχύει, ισχύει και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε για παραπάνω, παραπάνω γραπτά. Αν θέλετε, η Καβριέλα σημειώνει και ευχαρίστω γραπτά να σα στείλω περισσότερε πληροφορίε. Κύριε Όγκεν τώρα. Ένα τρίτο των χωρών μελών λέμε. Λέτε ότι είναι δύσκολο ακόμα και έξι χώρε να μπορέσουν να έχουν μια κοινή πρωτοβουλία. Εντάξει, σα πιστεύω. Αλλά από την άλλη, οι έξι χώρε μέλη, οι πολίτε αυτών των έξι χωρών, θα προτείνουν μια νομοθεσία που θα πρέπει και 27 μετά να εφαρμόσουν. Γι' αυτό και είμαστε διστακτικοί να συμφωνήσουμε για χαμηλότερο αριθμό χωρών. Γιατί τότε δεν είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αυτή. Την προτείνουν 6 χώρες και θα πρέπει να την εφαρμόσουν 27. Εκτός μικροφώνου παρεμβαστής κ. Ρόγκαν. Ναι, όντως από την αρχή υπήρχε πρόταση του ενός τρίτου. Για την ηλικία των 16 ετών και ότι θα φτάσουν 18 μέχρι να έχει προχωρήσει κάτι. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, σε αυτό συμφωνώ μαζί σας ότι συνήθως παίρνει χρόνο, παίρνει χρόνο να ολοκληρωθεί μια διαδικασία νομοθετικής πράξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξανασυζητηθεί πάντως αυτό το θέμα με τα κράτη-μέλη, έτσι κι αλλιώς στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Αυτό που είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποφεληθεί για να αποκτήσει περισσότερη δημοτικότητα, συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, γιατί το νόμο για την Ισπανία και τις ακτές εκεί. Είναι πολύ δική η ερώτησή σας. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω αρκετές πληροφορίες γι' αυτό. δεν είναι ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η ιδιοκτησία. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα θέλετε να ετοιμάσω κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά να σας το δώσω γραπτά, γιατί δεν έχω μαζί μου ό,τι χρειάζομαι για να σας απαντήσω. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση στην ενημέρωση, ξέρετε ότι έχουμε συνεχιζόμενες διαδικασίες για το 1049, πρόσβαση δηλαδή στην ενημέρωση, είναι οδηγία 1049. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρουμε ότι πιέζει προς μία κατεύθυνση, τα κράτη-μέλη πιέζουν προς μία εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και η Επιτροπή προσπαθεί να συμβιβάσει αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Το χάσμα όμως είναι τόσο μεγάλο που μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουμε κάτι. αν η πρώτη ανάγνωση και οι τροπολογίες δεν εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πάντως που θα μας βοηθούσε θα ήταν αν επικεντρωνόσασταν στην πρόσβαση στην ενημέρωση για τους πολίτες και να μην μπαίνατε σε λεπτομέρειες για το τι κάνουμε με τις απόρριτες, τις χαρακτηρισμένες απόρριτες δηλαδή. Όχι. Χτες με τα διαμεσολαβητή και συζητήσαμε το πόρταλ, συζητήσαμε πώς μπορούμε να έχουμε για τους πολίτες κάποιους προσανατολισμούς σε πιο εύκολη μορφή. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε την νέα πύλη, το νέο πόρταλ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν αλλά δεν είναι γνωστές συχνά. Χτες λοιπόν μίλησα και με τον επικεφαλής του γραφείου του διαμεσολαβητή και από ό,τι κατάλαβα μετά τη χθεσινή συζήτηση, εντυπωσιάστηκα γιατί η πύλη αυτή είναι υψηλή ποιότητα. Αν έχουμε κάτι τόσο καλό, να το χρησιμοποιούμε, να το δείχνουμε στους πολίτες μας, ώστε να το χρησιμοποιούν πιο συχνά. Κύριε Χέφνερ, νομίζω ότι σας απάντησα για το θέμα του παραδεκτού. Συμμετείχατε και εσείς στη συζήτηση, οπότε το ξέρετε ότι προσπαθούμε να βρούμε από κοινού μια λύση. Απάντησα και για τις ταυτότητες, τους αριθμούς ταυτότητας, τα στοιχεία. Και εδώ θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση που να μπορείτε να δεχτείτε και εσείς και τα κράτη-μέλη. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Έχουμε ένα χρόνο για online συλλογή και θέλετε να έχουμε περισσότερο από ένα χρόνο αν δεν είναι online η συλλογή υπογραφών. Έτσι δεν είναι, αν είναι με χαρτί. Γραπτά. Καλά, πρέπει να το δούμε. Και για τις ακροάσεις συμφωνώ μαζί σας. Να δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Τώρα για την διαδικασία επιπαραβάση. Για τις διαδικασίες αυτές. Δεν είναι μυστικό ότι δεν είσαστε η μόνη επιτροπή που ενδιαφέρεται για την διαδικασία επιπαραβάση Όταν πρόκειται για διαδικασία επιπαραβάση για εμπορικά ζητήματα είναι η Επιτροπή για το εμπόριο που ενδιαφέρεται και αντίστοιχα η κάθε Επιτροπή. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό για όλους μας είναι να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία να ενσωματώνεται ορθά στην εθνική νομοθεσία και να υπάρχει πάντα τρόπος διόρθωσης. Χρειάζεται συνεργασία στον τομέα αυτό για να υπάρχει βελτίωση. Έχουμε διαπραγματεύσει με την ομάδα εργασίας σας όσον αφορά την ε, συμφωνία πλαίσιο. Ελπίζω ότι θα στηριχτεί η συμφωνία πλαίσιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά σας πολύ σύντομα. Συμφωνούμε ότι επιπλέον από ειδικέ και αιτήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή Τη κοινοτική νομοθεσίας, θα φροντίσει η Επιτροπή να δώσει πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις διαδικασίες επί παραβάση, ακόμα και κατά περίπτωση εφόσον το ζητεί το Κοινοβούλιο και τηρώντα βέβαια το απόρριτο έτσι όπως το έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάθε φορά που έχουμε μια διαδικασία παραβάση. Μπορείτε να δείτε λοιπόν όλες τις πληροφορίες, ποιες περιπτώσεις βρίσκονται στη διαδικασία επί παραβάση. Επίσης, εφόσον σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μία ή η άλλη ε, περίπτωση, ευχαρίστως να σας δώσουμε και πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Συγχρόνως όμως πρέπει να σας πω ότι πρέπει να τηρούμε και την ομολογία και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας και τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επί παραβάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι κι αλλιώς προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση για το κράτος μέλος, έτσι ώστε να την αποφύγουμε αυτήν τη διαδικασία επί παραβάση, να την προλάβουμε. Προσπαθούμε τα κράτη-μέλη να διορθώνουν τη στάση τους πριν φτάσουμε στην εφαρμογή της διαδικασίας επί παραβάση. Υπάρχει δηλαδή μία διαβούλευση πριν από τη διαδικασία επί παραβάση. Και όταν υπάρξει η διαδικασία και προχωρήσει, φροντίζουμε και πάλι να βρούμε τρόπους συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο πολύ, αλλά μου κάνατε πολλές ερωτήσεις. Τι να κάνω και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που δείξατε να με ακούσετε. Σας ευχαριστώ και εγώ και ζητώ συγγνώμη γιατί όντως σας υποβάλαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ και νομίζω ότι μπορούμε να διακόψουμε εδώ την συνάντηση με τον κύριο Σεύκοβιτς. Αφού ευχαριστήσαμε τον Επίτροπο Σεύκοβιτς, θα θέλουμε να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη και μετά από την αλλαγή που είπαμε θα έχουμε, θα πάμε στο σημείο 10 την αναφορά του Αλμπέρτο Περίνο, εξονόμας της Ένωσης Habitat, σχετικά με την αντίθεσή του στην υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής δρομικής γραμμής ψηλής ταχύτητας μεταξύ των πόλεων Τωρίνο και Λιών και επίσης Μάρκο Τομαλίνο και Παύλο Πριέρη και τον Ρέμο Καστανιέρη και Αλμπέρτο Παύλο Βέτζο. Είναι στο 10 όλες αυτές είναι παρόντες. Ε, ξεκινάμε από τον Αλμπέρτο Περίνο, ο οποίος και θα λάβει το λόγο. Απόν ο κύριος Αλμπέρτο Περίνο για το σχέδιο κατασκευής δρομικής γραμμής μεταξύ των πόλεων Τωρίνο και Λιών. Perfetto, quindi allora Δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί ο κύριος Αλμπέρτο Περίνο. Ο κύριος Πάολο Πριέρη έχει τον λόγο, ο οποίος εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο και τον κύριο Αλμπέρτο Περίνο. Εντάξει, θα πάρετε και το έγγραφο, μπορείτε να λάβετε τον λόγο πάντως εσείς. Ο κύριος Πάολο Πριέρη. There Κάποιος που θα ήθελε να λάβει το λόγο να βοηθήσει. Okay. Αυτά. Μέχρι να μας έρθει και ο τεχνικός για να κατεβάσει την οθόνη ή όχι. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ζητήσω από την πρόεδρο να μπορέσω να διαβάσω μια σύντομη ευχαριστία. Εντάξει, εντάξει, αλλά σας παρακαλώ σας παρακαλώ. Και αυτό προς το συμφέρον σας ε, όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί τα έχουμε διαβάσει αυτά. Διαφορετικά θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους της Επιτροπής για να δούμε και μια δεχόμενη απόφαση. Λοιπόν, ε, καλημέρα σε όλους, εξ ονόματος των πολιτών στο Νόταβ που εδώ και 21 χρόνια είναι κατά της νέας αυτής σύνδεση, ε, μεταξύ των δύο πόλων γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να σας δώσουμε πληροφορίες ε, φρέσκε, φρέσκες, ενημερωμένες για την κατάσταση σημερινή κοινωνική πολιτική αυτών των περιοχών που διασχίζει η γραμμή αυτή και έτσι ε, θα δώσουμε ταυτόχρονα και ορισμένα έγγραφα στην Επιτροπή Αναφόρων και θα απαντήσουμε ευχαρίστω στα ερωτήματά σα. Μια σύντομη εισαγωγή γενικού χαρακτήρα. Οι Ιταλοί πολίτε που εξονόματο πολλών επιτροπών ε, στα πλαίσια τη κίνηση Νοτάβα ανάμεσα στο 2003 και 2008 επέδωσαν έξι αναφορέ και ελπίζουμε, περιμένουμε να λάβετε κατάλληλε πρωτοβουλίε ε, ώστε να διαβαστούν προσεκτικά αλλά υπάρξουν και απαντήσει χωρίς καθυστέρηση να δείξει ότι είναι πραγματικά ε, οι ευρωβουλευτές πολιτικά υπεύθυνοι και όχι μόνο την απάντηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά θέλουμε να ξέρουμε, ε, θέλουμε να καταλάβουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίζει αυτόνομο ρόλο απέναντι στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια δεν αναφέρεται, δεν λαμβάνει υπόψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα δικαιώματα των ατόμων αλλά τα δικαιώματα των ομάδων πίεσης και ε, θα σας πούμε ότι με ανεξάρτητα όργανα, με ανεξάρτητους πανεπιστημιακούς να μπορέσουμε να έχουμε γνωμοδοτήσεις μετά από όλα αυτά που εξετάζουμε το μανιφέστο το ευρωπαϊκό για τα τρένα υψηλή ταχύτητα, μια πραγματική δημοκρατική ενιαία συζήτηση για τα πρότυπα μεταφορά, για την ανάπτυξη επιτόπου, κοινωνική και για να μην πραγματοποιηθούν αυτά σχέδια υποδομής και λοιπά που είναι, γίνονται μετά από πίεση των λόμπις. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Και τώρα την απάντηση του Αλμπέρτο Περίνο για την 949 αναφορά, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα γραμμή από 21 χρόνια και μετά οι κάτοικοι, οι τεχνικοί όλοι είναι κατά αυτού του έργου. Αυτό έχει μια σημασία, ένα νόημα πριν από πολλά χρόνια ξεκίνησαν τη συζήτηση για αυτή την σύνδεση και με πάρα πολλά τούνελ και τότε φτιαχνόταν και ο δρόμος Α32 που για πάρα πολλά χρόνια χαλούσαν τη ζωή των κατοίκων εκεί και χάλασαν και το περιβάλλον εκεί στις κοιλάδες αυτές καταλάβαιναν ε, κατάλαβε ο κόσμος τι θα σήμαιναν άλλα 30 χρόνια προβλημάτων, ε, ε, προβολική κίνηση, δύσκολη επικοινωνία και όλα αυτά μαζί με τους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και λοιπά λοιπόν. Επίσης στο Στρασβούργο πήγε μια αντιπροσωπεία δική μας ε, και επέδωσε στο πρόεδρο του Κοινοβουλίου μια επιστολή με 32.000 υπογραφές που ενδιέφερε αυτή η νέα γραμμή του Ρήνου Λιών και όχι μόνο. Οκτώ, οκτώ τόμοι υπογραφών ε, ότι ήταν αντίθετη και ότι η κοιλάδα της Σούζα δεν μπορούσε να δεχτεί παρόμοιο έργο. Τις 10 Αυγούστου του 2010 και έγινε γνωστό το προκαταρτικό σχέδιο για το κοινό μέρος της νέας αυτής συνδρομικής γραμμής. Από Ιταλικής πλευράς δεν ακούστηκε τίποτα συγκεκριμένο γιατί δεν παρουσίασε ούτε το προκαταρτικό σχέδιο ε, ο Ιταλικός ιδερόδρομος αλλά θα ήταν κάτι καταστροφικό οικονομικά, περιβαλλοντικά και ο Υπουργό Τρεμόπτη είπε θα είχε τρομερό υψηλό κόστος και προς το παρόν ε, υπάρχει μόνο το ξεκίνημα ενός τούνελ. Πολλά υποσχέθηκε η Ιταλική κυβέρνηση, αλλά δεν έκανε τίποτα, δεν έχει χρήματα για να επενδύσει και τις 17 Σεπτεμβρίου σε μια συγκέντρωση από τους βιομήχανους του Πεδεμοντίου ο κύριος Σινιόρε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ΕΛΚ, δήλωσε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα για παιδικούς σταθμούς ε, είναι δίκαιο να ξοδευτούν 20 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα έργο παρόμοιο που όπως μας προτείνεται δυστυχώς θα καθυστερήσει πάρα πάρα πολύ σε σχέση με την οργάνωση και όλα αυτά θα έχει τρομερό κόστος και ουσιαστικά θα εξυπηρετεί μόνο για τους επιβάτες και θα ξοδέψει, θα σπασταλίσει χρήματα μια κάποια στιγμή που χρειάζονται αυτά χρήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραμείνουμε σιωπηλοί. Και στην κοιλάδα της Σούζο παρά το κίνδυνο αυτό οι τεχνικοί, οι διοικητικοί υπάλληλοι εξέτασαν αυτά τα προγράμματα και ε, ξετρελάθηκαν όταν άκουσαν αυτά τα πράγματα και υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι και πραγματικά θα ήταν και εις βάρος της υγείας των πολιτών για υπερευαίσθητες σε καρδιογιακά προβλήματα ε, μερίδες πληθυσμού, ο αμίαντος κλπ. Και ταυτόχρονα πολλά βράχια που ίσως είναι μολυσμένα και που θα μολύνουν τον ε, χώρο με και τον αέρα με την σειρά τους. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Και ο νομοθέτης ε, είπε ότι ο αμύαντος δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε παραμικρή υποψία για την άνοιγμα αυτών των ε, τούνελ. Επίσης θα επηρεάσει το νερό ε, στο τούνελ αυτό και αυτό είχε δειχτεί από ένα έγγραφο, μια ανάλυση από την ETF, από το αρμόδιο οργανισμό και από, με την κυρία Ντεπαλάθιο. Και τώρα στο σχέδιο αυτό αναφέρεται ότι ε, στην έξοδο θα έχουμε εντάξει μια ισορροπία, θα έχουμε 1040 όμως λίτρα νερό που θα χάνονται, πάρα πολλά κυβικά καθημερινά και εκεί δεν υπάρχουν γεωλογικά στοιχεία και τότε ανάμεσα θα δίνουν περίπου 60.000 κυβικά μέτρα το μέρα που θα χάνονται. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τον Ούρε στο Μουτζέλο που συνέβη ένα ατύχημα και τότε ξεράθηκε ε, μια ε, ξεράθηκαν, στέρεψαν 37 πηγές και η ζημιά ήταν 740 εκατομμύρια περίπου ευρώ, τόσο υπολογίστηκε. Επίσης ε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται να φτιάχνει ένα παρόμοιο έργο είναι ασύμβατο, ε, είναι απαράδεκτο, έχει τρομερό κόστος ε, παρόλη την συμβολή τη γαλλική και την ιταλική και όπως είπε και το παρατηρητήριο υπό τον κύριο Βιράνο και να υπενθυμίσουμε ότι η σημερινή γραμμή εξυγχρονίστηκε τώρα τελευταία ανάμεσα στη Λιόν και στο Τωρίνο και το Δεκέμβριο φέτος θα περατωθεί το γαλλικό μέρος και θα έχουμε βέβαια ε, τρένα υψηλής ταχύτητας για τους ε, επιβάτες, αλλά πέσαμε στα επίπεδα του 50 για τα εμπορεύματα. Θα πρέπει να διακοπούν ε, οι, τα κονδύλια, η χορήγησή τους για αυτό το έργο, για να μην καταστραφεί το περιβάλλον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το LCA, Life Cycle Assessment, για το σύνολο του σχεδίου αυτού και σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Αλμπέρτο Παολοβέζιο. Eh, Σας ευχαριστώ και χαιρετώ όλους. Έχει να κάνει έκθεση η αναφορά αυτή με το ότι η διοίκηση η τοπική και ο τοπικό πληθυσμό δεν συμμερίζονται πουδενή τι διάφορες φάσει τη προκαταρτική του σχεδίου και τώρα το σύνολό του. Έχουμε διάφορα στοιχεία βέβαια σίγουρα συγκεκριμένα που δείχνουν ότι δεν είναι σύμφωνος ο ντόπιο πληθυσμός και το παρατήριο εκεί που συμμετέχει και η τοπική αυτή δεν είναι κάτι το αντεσπευτικό γιατί έχουμε δύο μόνο από ό,τι βλέπουμε στην διαφάνεια δύο μόνο από όσους ενδιαφέρονται και συμμετέχουν σε αυτό και υπάρχουν δεκάδες δήμοι που δεν τους ενδιαφέρει το έργο αυτό. Στα πράσινα και στα κόκκινα γραμμή βλέπετε την γραμμή αυτή τη συνδρομική και δεν είναι κανονικό όλοι αυτοί οι δήμοι που δεν τους αφορά το θέμα παρόλα αυτά συμμετέχουν στο παρατηρητήριο. Όπως και στο παρελθόν και τώρα δεκάδες δήμοι και πάλι αποφασίζουν κατά της γραμμής αυτής. Το 2008 εδώ στο Κοινοβούλιο ε, δόθηκαν αναφορές και υπογραφές από δεκάδες φορείς που ήταν αντίθετοι με αυτό το έργο. Και εδώ με το κόκκινο βλέπετε όλους τους Δήμους που στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν εξ αυτήν την απόψή τους κατά, κατά του έργου αυτού. Βλέπετε την μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη ναι του παρατηρίου και στα όσα λέει ο κόσμος. Και επίσης και άλλοι. Υπάρχει ένα έγγραφο, ένα έγγραφο που αναφέρθηκε και από την Επιτροπή σας σε μια απάντηση ενδιάμεση που δόθηκε στην αναφορά μας. Το σχετικό έγγραφο είναι μόνο μια περίληψη αυτό που είχε αποφασίσει ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου για το πώς θα έπρεπε να χαραχθεί η γραμμή. Και μόνο εκείνος το υπέγραψε. Βλέπετε αυτό το θέμα, αυτό κάτω-κάτω εκεί τη συμφωνία, την υπογραφή και την υποσημείωση. Κανονικά θα πρέπει να υπογραφεί από όλου και από τον προτείνοντα και από τους υπόλοιπους. Εμείς σαν αύριο το πρωί να λέγαμε ότι εντάξει συντάσσουμε ένα έγγραφο που να λέμε συμφωνία των Βρυξελών, να βάλουμε όλα αυτά, ότι θα πρέπει να αναχαιτιστεί, να παγώσει κλπ. Το υπογράφαμε εμείς και μετά το παρουσιάζαμε στους ε, δημοσιογράφους και λέγαμε ότι όλη η Επιτροπή, το σύνολο της Επιτροπής Αναφορών ε, συμφωνεί. Άρα λοιπόν θα ήταν κάτι ψεύτικο. Κάτι τέτοιο συνέβη με την απόφαση εισαγωγικά του παρατηρητηρίου. Και ακόμα μια δεύτερη πτυχή που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι δεν συμφωνεί ο ντόπιο πληθυσμό ε, που βασίζονται όλα αυτά σε τρία ε, εκφράζονται με τρία, βασικά στοιχεία. Πρώτα 20 χρόνια, ε, τρία, τρία χρόνια ουσιαστικά, 20 ε, χρόνια ε, σχεδιάζεται αυτό το έργο, αντιδρά ο πληθυσμό και ουσιαστικά έχει δοθεί ε, χαρακτήρα στρατιωτικής επιβολής εκεί. Εδώ όλοι αυτοί που πάνε από τα σύνορα τα γαλλικά μέχρι το Τωρίνο συμμετέχει και μια επιτροπή αγώνα συμμετέχουν εκατοντάδες άτομα και χιλιάδες άτομα και ε, βραδιές ενημερωτικές οργανώθηκαν και βλέπουμε ότι δίδονται και πολλά κονδύλια από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σπαταλιούνται. Εδώ εμείς προβλέψαμε ε, και στην Όλαφ ε, για τις απάτες και τα σταλίες να καταθέσουμε αναφορά. Και βλέπουμε ότι και, στο μέλλον τον 1 Οκτωβρίου θα γίνει μια πορεία όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι Δήμοι και χιλιάδες πολιτών. Και το παρατηρητήριο βλέπουμε ότι δίνει ψεύτικα στοιχεία και εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό και από τα χειρότερα που δείχνουν τη διάθεση ε, να επιμείνουν σε αυτές τις αποφάσεις ε, του παρατηρίου. Ε, βλέπουμε όμως ότι και το, ε, και το παράρτημα 1 παραβιάζεται που επικυρώθηκε και από την Ιταλική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες σε αποφάσεις αφού γνωρίζουν πρώτα το θέμα αλλά και την απόφαση του δικαστηρίου που λέει για την εγγύηση της πρόσβασης της πληροφορίες. Αυτό δεν ε, έγινε σεβαστό και δεν φαίνεται καλά ίσως από τον αδιαφάνεια αλλά αριστερά βλέπετε στο περιφερειακό ε, Διοικητικό Δικαστήριο του Παιδεμαντίου, του Τωρίνου, φαίνεται η απόφαση. Ε, βλέπουμε ότι το παρατηρητήριο αποδεικνύεται ότι δεν μας παραχώρησε πρόσβαση στα έγγραφα και καταδικάστηκε ουσιαστικά το παρατηρητήριο αυτό ε, γιατί δεν επέτρεψε δική μας πρόσβαση των στοιχείων. Η απόφαση αυτή του Ιουλίου του 2008 δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Και εμείς βέβαια πώς το πω τώρα, εμείς εξοδικαστικά εδώ δίπλα ε, βλέπετε πώς προχωρήσαμε για να ε, υπάρξει κάτω εγγυημένο σαν πρόσβαση, ότι και αυτό είναι σεβαστό και τώρα εμείς ετοιμάζουμε ε, μια κατάλληλη ενέργεια για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε το σημείο αυτό, γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερα δεινό, το κάτι το αρνητικό. Θα πρέπει να σεβαστεί την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, το παρατηρητήριο. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα που σα είπα τώρα, ότι δεν σέβονται, δεν υπάρχουν συνθήκε και όλα αυτά. Εκτό από το ότι αυτά τα εγγραφά που λένε για την γραμμή, ότι πρέπει να γίνει, αυτά τα επιχειρήματα είναι συχνά από διοικητική οικονομικής πλευράς. Εδώ ένας άλλος λόγος είναι ότι διατηρώντα μυστικά όλα τα υπόλοιπα, οι πολίτε έτσι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση πώ δαπανώνται. Παράδειγμα, έτσι, ένα τυχαίο γεγονός, μόνο τυχαία μάλλον, ε, καταλάβαμε, είδαμε στοιχεία πώς η LTF, αυτή η εταιρεία για τις φυγομετρήσεις, πλήρωσε σε μια άλλη εταιρεία που στο χώρο της θα γινόταν ε, αυτή η σφυγομέτρηση, πλήρωσε 160.000 ευρώ για δύο περιοχές για την ενοικίαση ε, για 11 μέρες αυτά τα 160.000 ευρώ είναι τρομερό ποσό. Ε, άλλωστε και γι' αυτό προσφύγαμε στην ε, υπηρεσία κατά της απάτης ε, Όλαφ και παρουσιάσαμε, υποβάλαμε το εγγραφό αυτό με την απόδειξη αυτή και στην Ιταλία και βλέπουμε ότι υπάρχει 667 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Η Ιταλική κυβέρνηση πλήρωσε 35.000 ευρώ ε, για έξοδα ξενοδοχείων για την αστυνομία που θα προστάτευε το χώρο για να ε, χαραχθεί το έργο. Εδώ λοιπόν ε, ζητάμε αυτά τα 678 εκατομμύρια να παγώσει η παραχώρησή τους μέχρι να γίνει με ένας έλεγχος του λόγου ε, κόστους οφέλους και να δούμε ε, το πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, τι έγινε, πώς έκαναν αυτές τις παραχώρησεις οι διεθνείς πιέσεις. Να δούμε και την απόφαση, γιατί δεν δείχνει καθαρά ε, ποια είναι αυτή η δαπάνη, πώς έχει, τι γίνονται αυτά τα χρήματα. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, μάλλον η εκπρόσωπος Επιτροπής Κατρίν Πρίντς. Ε, well, uh, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που δίνετε το λόγο στην Επιτροπή. Έχουμε απαντήσει σε αυτές τις αναφορές και γραπτός. Περιληπτικά, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την διαδρομή αυτή που ξεκινάει από την Λιό και φτάνει στην Ουκρανία, πρόκειται για ένα σχέδιο με προτεραιότητα, κάτι το οποίο επιβεβαιώσαμε το 2004, κάτι που βεβαίως μπορεί να εξηγηθεί με μια πολύ σημαντική μελέτη που έγινε σε μια περιοχή από περιβαλλοντολογικής απόψεως εξαιρετικά ευαίσθητη, η περιοχή των Άλπαιων, η σημερινή κυκλοφορία που περνάει από τη Λιόν προς το Τωρίνο είναι μια διαδρομή με όλες ε, τις ε, αν θέλετε, μειονεκτικές πλευρές μιας διαδρομής η οποία υπάρχει εδώ και αιώνες και η οποία έχει δείξει τις δυσκολίες της σήμερα η σύραγγα που υπάρχει εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια και έχει τελειοποιηθεί όσον αφορά την Ιταλική της ε, πλευρά, πρέπει να τελειώσει η Γαλλική πλευρά, συνεχίζει και ε, έχει κάποια μειονεκτήματα. Παραδείγματο χάρη αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να υπάρξει κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας η πρώτη μελέτη που έγινε στο τέλος Νοεμβρίου του 2005 από την Αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την μεταφορά όλων αυτών των, όλης αυτής της κυκλοφορίας από τους δρόμους, από τις ειδικές μεταφορές, τους σιδηροδρόμους, έδειξε στα πορίσματά της ότι χρειαζόταν περαιτέρω μελέτη. Ο ε, συντονιστής, ο Ευρωπαίος συντονιστής, συναντήθηκε με όλους τους κοινωνικούς ε, φορείς, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αύριο υπάρχει μια άλλη συνάντηση έτσι ώστε να λυθούν όλα αυτά τα σημεία υπόψη για το μέλλον η χρηματοδότηση, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά και η γαλλική και η τελική χρηματοδότηση βασίστηκε σε μελέτες. Μελέτες των οποίων ο αρχικός στόχος ήταν να δούμε εάν υπάρχουν περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις και να βρεθεί τρόπος να καλυφθούν, να εξουδετερωθούν ε, ή να εξαλειφθούν τελείως αυτές οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Ακούω από τους αναφέροντες ότι υπήρξαν εβδομαδιαίες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους εκπροσώπους των Δήμων, όλους τους Δήμους που ήθελαν να εκπροσωπηθούν. Αυτές οι συναντήσεις μας οδήγησαν στην αλλαγή κάποιων τμήματων αυτής της διαδρομής, ιδιαίτερα μια πολύ αμφισβητούμενη και προβληματική περιοχή στο Βενάους. Συμμορφωθήκαμε λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των τοπικών κοινοτήτων και φορέων και είδαμε ότι αυτή η νέα διαδρομή υποστηριζόταν από τους περισσότερους. Προσπαθήσαμε επίσης να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες. Βεβαίως, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες εξκαφές για την εξέταση του εδάφους, της ποιότητας του εδάφους, ε, ελήφθησαν υπόψη οι προδιαγραφές για τέτοια έργα, όπως γίνεται πάντοτε. Σας ευχαριστώ. Κάποιος συνάδελφος που θα ήθελα να λάβει το λόγο. Όκεν. Sorry, sorry. Yeah. I'm really tired now. Ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να ζητήσω κάτι από την Επιτροπή. Περιγράφεται αυτή την διαδρομή, την παλιά διαδρομή. Ναι, υπάρχει. Μιλάμε για εξυγχρονισμό και αυτή η ανοικοδόμηση ή όπως θέλετε μπορείτε να την ονομάσετε, αναπροσαρμογή μιας παλιάς ε, διαδρομής, σίγουρα έχει πολύ λιγότερες συνέπειες από αυτή της δημιουργίας μιας σύραγγας εκ νέου από το τίποτα. Και τελικά έχει γίνει η μελέτη για το ποιος θα επωφεληθεί Ποιο θα χρησιμοποιήσει πραγματικά αυτή τη νέα σύραγγα. Η έκθεση περιβαντολογικών ε, επιπτώσεων έγινε. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ζητάμε και έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε σαφή απάντηση και αυτό με εκπλήσει υπάρχουσα διαδρομή γιατί δεν βελτιώθηκε, εξυγχρονίστηκε. Μιλάμε για τα τρένα υψηλής ταχύτητας που φτάνουν τα 380 χιλιόμετρα την ώρα. Μα ποιος χρησιμοποιεί αυτά τα τρένα. Ποιος τα χρειάζεται. Οι παραδοσιακές γραμμές μπορούν να βελτιωθούν και ίσως αυτό ήταν το ζητούμενο. Συνάδελφος Κάντσαν. Ναι, να πω κάτι προκαταρτικό σημαντικό. Είμαι υπέρ μια διαφάνεια τη προκήρυξη διαγωνισμών και αυτό για την προστασία του περιβάλλοντο, για τι προδιαγραφέ, τι καλύτερε τεχνικέ πρακτικέ, όλα αυτά. θα πρέπει να κρατήσουμε σταθερή θέση οπωσδήποτε απέναντι στα τέσσερα αυτά σημεία που αποτελούν και τις αρχές μας για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα, για την πρακτική εφαρμογή αυτών των αρχών και για να παγώσει η κατασκευή αυτού του διαδρόμου που θεωρείται σημαντικότατο στην Ευρώπη. Τώρα, χρειάζεται να το σκεφτούμε αρκετά. Στην Επιτροπή μου Μεταφορών ομόφωνα εκφράστηκε η άποψη ότι ε, θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος μεταφοράς όχι πια οδικά αλλά σιδηροδρομικά. Και για το μέλλον έχει σημασία αυτά. Θα είναι από τους, το έξι αυτός ο σημαντικότατος διάδρομος που οριζόντια συνενώνει την Ανατολή με τη Δύση, την κυκλοφορία, την οικονομία. Τώρα να το κόψουμε αυτό το κομμάτι επειδή δεν συμφωνούμε το πώς, με ποιο τρόπο, τι να πω τώρα περισσότερο, δεν θα πω κάτι παραπάνω γιατί ε, ίσως δεν είμαι και τόσο γνώστης του θέματος. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαστε εμείς που να διακόψουμε την κατασκευή αυτού του διαδρόμου. Όταν λέμε ότι τα τρένα ψηλής ταχύτητας ε, είναι απαραίτητα, αυτό αποτελεί μία απάντηση έτσι σκέτη που απαιτείται καθαρή. Και εγώ λέω ναι, γιατί στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει αυτό το σύστημα τρένεψης ταχύτητας που είναι απαραίτητο και δεν θα ήθελα να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα σε αυτό το διάδρομο, σε αυτόν τον άξονα που πέρα από τις Αλπις να μιλήσω για την Ιταλία και εγωιστικά να πω ότι για τη χώρα μου την Ιταλία απαιτείται μια παρόμοια γραμμή. Γιατί, αν αυτό γινόταν μόνο από την άλλη μελεριά των Άλπαιων, τότε το πρόβλημα για αυτό το μέρος της Ευρώπης στην Ιταλία το βόλμα θα ήταν μεγάλο. Γι' αυτό για τον Επίτροπο Μπρίνχορστ θα ήθελα να τον παρακαλέσω. Ξέρω ότι προσέχει τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να τον παροτρύνω να μπορέσει να βρει την καλύτερη πρακτική, τις καλύτερες συνθήκες, να ισχύσουν οι καλύτερες προδιαγραφές, αλλά σας συγκετεύω δεν θα πρέπει να χάσουμε τη χρηματοδότηση αυτή για την κατασκευή του έργου, δεν θα πρέπει να παγώσει αυτό το έργο, γιατί σημαίνει ότι καταστρέφει τη δυνατότητα σύνδεσης βάσει του βασικού άξονα PP6. Κάποια άλλη παρέμβαση, όχι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι για την Επιτροπή. Όσα σήμερα αναφέρθηκαν από τον ε, σύμβουλο Πρινς δεν φέρνει κανένα στοιχείο καινούριο στην απάντηση επιτροπή αυτό που είχαμε από το Σεπτέμβριο του 2009. Δεν έχουμε καινούργια στοιχεία, σχεδόν τίποτα. Από το 2009 έλεγε ακριβώς η Επιτροπή ότι είχε παρακολουθήσει Κάμψη, δύσκολα σημεία, ότι είχε κάνει ελέγχους, ότι είχε δείξει ότι χρειαζόταν όπως και σε παρόμοιες παλιότερες φάσεις διαβουλεύσεις έγιναν αυτές, υπήρξαν διάφορες θέσεις και αντιπαραθέσεις. Σεπτέμβριο του 2009 λέει ότι δεν υπάρχει μια εκτίμηση σχετικά με τις παρεμβαλλοντικές επιπτώσεις. Ούτε σήμερα ακούσαμε κάτι τέτοιο. Τώρα, δεν ακούσαμε ούτε μια ελάχιστη απάντηση για αυτά που λένε οι αναφέροντες από ποιους αποτελείται ε, αυτό το παρατηρητήριο μέχρι το 2006 και μετά έχουμε τα διάφορα στοιχεία που αναφέρονται αλλά δεν είπε κανείς αν αυτό το παρατηρητήριο εκπροσωπεί πραγματικά ε, τις ανάγκες μιας σωστής συμμετοχής ε, της πληθυσμιακής βάσης όπως ακούσαμε από τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αυτό. Τι γίνεται με αυτό το πάγωμα των κονδυλίων που εξαρτάται από τον έλεγχο που προχωράει αν αυτοί, αυτές οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, σωστά, τακτικά ή μήπως μπαίνει για κάτι άλλο στη μέση που παρεμποδίζει. Um, Σας ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω καταρχήν σε αυτή την ερώτηση τότε. Δεν είπα τίποτα καινούριο από τότε που το 2009 απαντήσαμε γραπτός. Γιατί στην Ιταλία, ουσιαστικά επιτόπου, δεν συνέβη τίποτα καινούριο. Η έκθεση για τις περιβατολογικές ε, επιπτώσεις δεν ξεκίνησε ακόμα, γιατί δεν έχει δοθεί άδεια ακόμα για αυτήν την ε, πρώτη η τελική μελέτη στην Ιταλία. Γι' αυτό και δεν ξεκίνησε και το έργο. Όσον αφορά αυτό το παρατηρητήριο και την σύστασή του, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εβδομαδιαίες συναντήσεις ε, αυτού του παρατηρητηρίου, μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, τους σιδηροδρομικούς, τις περιφερειακές τοπικές αρχές. Βεβαίως, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμμετοχή. Κάποιοι έχουν επιλέξει να μην συμμετέχουν σε αυτό το παρατηρητήριο. Να απαντήσω σε κάτι που ρώτησε η συνάδελφό σας όσον αφορά την σύραγγα αυτή σαφώς και σήμερα αναβαθμίζεται έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν μεγαλύτερα τρένα. Όμως αυτή τη στιγμή δεν λύνονται όλα τα προβλήματα γιατί το πρόβλημα της ακαμψίας παραδείγματος χάρη και το θέμα του περάσματος από ορεινές περιοχές, τα προβλήματα με τη χειμερινή περίοδο και το ψύχος. Όπως ξέρετε, όλα αυτά δεν μπορούν να ξεπεραστούν και η υπάρχουσα διαδρομή να καλύψει όλα τα προβλήματα και να περάσουν παραδείγματο χάρη τρένα υψηλής ταχύτητας. Απαντώ ε, εγώ στην στο τμήμα μου και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι είπα και πριν, ε, θα έλεγα και τώρα, γιατί είμαστε στην ίδια κατάσταση. Η οδηγία είναι διαδικασία ε, οδηγία εκείνη για τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος. Και η απόφαση λαμβάνεται μετά από τη διαδικασία. Αν κάποιος θέλει να φτιάξει στη Βιά τη Αναβόνα στη Ρώμα ένα πυρηνικό σταθμό, μπορεί να το κάνει ακόμα και αν φανεί ότι αυτό είναι αδύνατον. Γιατί, Γιατί είναι δύο διαδικασίες διαφορετικές. Άλλη η απόφαση και άλλη η διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ισχύει, όπως και στην 11 ότι δηλαδή υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην Ιταλία και την Σλοβενία ή την Ιταλία και την Γαλλία. Εμείς θέλουμε φυσικά τις βέλτιστες πρακτικές και είναι καλό αυτό που ακούσαμε σήμερα από τους αναφέροντες. Ευχαριστώ. Sí. Ε, ένα λεπτό απάντηση, όχι περισσότερο, έτσι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρώτα η... Θα θέλετε να λάβετε λόγο. Πολύ σύντομη ερώτηση. Ίσως έχετε δίκιο ότι η έκθεση για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν ξεκινήσει το έργο και τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Όμως, οι απαντήσεις της Επιτροπής είναι διαρκώς ίδιες. Αυτό δεν έχει νόημα. Μας λέτε δεν υπάρχει απολύτως καμία επίδραση. Αυτό πραγματικά το θεωρώ κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε υπάρχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία που μας λένε ότι αυτό θα πρέπει να μας φοβίζει, αλλά όχι. Τουλάχιστον να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μια τέτοια διαδικασία σαφώς θα αύξανε την εμπιστοσύνη των πολιτών. This Έχουμε 25 χρόνια της οδηγίας και στην Λουβέννη υπό τη Βελγική Προεδρία έχουμε μια σχετική τελετή. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι είναι μια μοναδική οδηγία αυτή επιπτώσεων περιβαλλοντικών γιατί επιτρέπει διαβούλευση με το κοινό. Καμία άλλη οδηγία δεν είναι σαν κι αυτή. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο όφελος από την οδηγία. Γι' αυτό που λέτε, βέβαια έχετε δίκιο. Η Κομισιόν το γνωρίζει. Εμεί θέλουμε να είναι πιο δυνατή η οδηγία. Η πραγματικότητα όμω είναι αυτή που είναι. Υπάρχει Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και για μα είναι δύσκολο να αλλάξουμε τα πράγματα. Ξέρουμε τι λέτε, το καταλαβαίνουμε, το έχουμε υπόψη μα. Είναι σημαντική χρονιά αυτή. 25 χρόνια από την έναρξη τη οδηγία σα φροντίσουμε να την κάνουμε πιο δυνατή στο μέλλον. Θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικός. Λοιπόν, απάντηση για τις δυνατότητες της γραμμής της σημερινής. Για την εμπορική γραμμή. Τα μισά εμπορεύματα που περνάω από την Ιταλία προς τη Γαλλία και από την άλλη πλευρά προς τα δω, από ότι 20 χρόνια πριν 5 εκατομμύρια τόνοι, έτσι σίγουρα. Αλλά λοιπόν υπάρχει δυνατότητα Αυτά τα 5 εκατομμύρια που δείχνουν την κυκλοφορία εμπορευμάτων είναι το 1 τρίτο της δυνατότητας της γραμμής. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι σιδηρόδρομοι κρατικοί. Όταν μιλάει κανείς για τη δυνατότητα, εντάξει, αυτό για το μέγεθος σύραγγας, πολύ σωστά, γιατί νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από γαλλικής πλευράς. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό, επειδή είμαστε στο 1 τρίτο της δυνατότητας μεταφοράς. Κάτι ακόμα για το παρατηρητήριο. Είπα κάπως, το κάπως έτσι ακαδημαϊκά, διδακτικά. Εδώ, εντάξει, ε, όχι επειδή εμεί επιμένουμε, εσείς συμφωνείτε, εντάξει, μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 δεν ε, ίσχυε αυτό ότι συμμετείχαν οι Δήμοι στο παρατηρητήριο. Εγώ είδα όλες ε, τις επιστολές των Δημάρχων που έλεγαν ότι δεν είχαν ποτέ σχέση με το παρατηρητήριο. Αλλά ο Δήμος θα πρέπει να συμμετέχει όπως και εμείς ε, συμμετέχουμε εδώ σε εσά. Δεν είναι ότι συμμερίζεστε αυτό που λέμε εμεί, ούτε εμεί αυτό που λέτε εσεί. Άρα λοιπόν το να λέει κανεί, το να διαδίδει και να λέει αυτό που λέει το παρατηρητήριο αυτό που υποστηρίζει μόνο ο πρόεδρος του παρατηρίου να λέει ότι το υποστηρίζουν όλοι. Τι να σας πω, δεν δε πάει, δεν στέκει αυτό το πράγμα. Για το... Εδώ βλέπετε αυτό το, είδατε προηγουμένως αυτό το έγγραφο που υπέγραψε ο πρόεδρος του παρατηρίου, όχι η Δήμη. Παντού Όλοι υπογράφουν, όχι μόνο ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν ε, να διαλύσουμε αυτή την αμφιβολία. Να ε, εξηγήσετε μου τι γίνεται αν πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι το αντίθετο. Εντάξει υπάρχει ένας φορέας παρόν και δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια αποδοχή. Διαφορετικά μυθοποιείται αυτό το πράγμα και κάποιος ε, από τη στιγμή που παρουσιάζει ένα έγγραφο του πρατηρητηρίου και από το 70 άντε 50% των δήμων εντάξει θα το δεχτούμε αυτό ο πρόεδρος και τουλάχιστον 50%. Αλλά ε, δεν ξέρω, από τη στιγμή που εμπιστεύεστε έγγραφα που παρουσιάζει ένα άτομο που υπογράφει εξ ονόματος όλων, επιτρέψτε μας το πω ότι αυτό δεν ε, στέκει, δεν είναι αποτελεί πραγματικότητα. Εντάξει, εμείς, ε, ε ναι, λέμε ότι όποιος θέλει ας το προχωρήσει. Εμείς ε, ε, αυτό το έγγραφο σας το δείξαμε, το υπέγραψε μόνο το παρατηρητήριο. Όποιος λέει ότι εντάξει στο παρατηρητήριο εκεί συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς, να μας φέρει ένα στο έγγραφο που να έχουν υπογράψει τουλάχιστον το 50% των Δήμων και όχι μόνος του ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. δεν είναι πλήρης η απάντηση της Επιτροπής. Δυστυχώς θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα ακόμα, όπως έλεγε και η συνάδελφος Όκεν, εδώ και χρόνια το συζητάμε. Πάντως παραμένει κάτι το εκρεμές, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας φέρουν εδώ και οι υπογράφοντες τις αναφορές. Αυτά τα στοιχεία είτε είναι βάσιμα είτε όχι, αλλά δείχνουν όλα αυτά ε, σχετικά με τη διαδικασία και πως λέει η Επιτροπή ότι όλα πάνε καλά και προχωρούν. Εμείς παρ' αυτά ε, λέμε ότι κάτι δεν στέκει εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει σίγουρα να διατηρήσουμε ανοιχτό το θέμα ή αυτές τις αναφορές ε, που έχουν να κάνουν με το ίδιο θέμα και να περιμένουμε μια απάντηση πλήρη σχετικά με τη διαδικασία και για την πιστοποίηση και το άνοιγμα, το πράσινο φως από τη μεριά της Ιταλίας. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει αυτό προς το παρόν. Από τη στιγμή που συνεργονούν και οι συνεδάδελφοι, αυτή τη λύση δίνουμε προς το παρόν. Καμία αντίρρηση. Άρα λοιπόν και αυτό θα γίνει. Παραμένει άνοιχτο το θέμα των αναφορών αυτών και το θέμα της αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπογράφοντες. Παρακαλώ κάτι θα ήθελα θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε. Δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε όμως και οι πέντε μας ε, τις απαντήσεις μας ε, στις αναφορές. Εντάξει, θα τα έχετε και στην ιστοσελίδα μας και εσείς θα τα έχετε στα χέρια σας ε, και μπορείτε να στείλετε στη μεταφορά αναφορές και περιβάλλον να στείλετε αυτές αναφορές μας σας εξουσιοδοτούμε δεν υπάρχει πρόβλημα έτσι ε, όλα αυτά έτσι, μέσα σε λίγη ώρα δεν μπορούν να λυθούν ε, όπως εδώ. Σας ευχαριστούμε όμως για το ανοιχτό πνεύμα που επιδείξετε απέναντι στη δημοκρατία, στην ευγένεια, στον πολιτισμό και γαλήνια εγκαταλείπουμε την αίθουσα αυτή. Σίγουρα ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος για να αποδειχτεί η αλήθεια και όχι οι μυθοποιήσεις ε, στυλ παρατηρητηρίου. Αυτά. Στο τέλος θα σας δώσουμε εδώ στην έξοδο και το σχετικό έγγραφο, τις σχετικές αναφορές, απαντήσεις μάλλον. Το επόμενο τώρα, 900-2007 Τζανκάρλο Παστορούτη, τη Επιτροπής ΝΟΤΑΒ και άλλων επιτροπών που ενωδιώνται στο διάδρομο 5 σχετικά με τη θέση του στην Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για τον Συνδρομικό Άξονα ταιριέ στην Τιβάτσα. Ο υπογράφων Απών. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν, ε, δεν μου το είχαν πει. Ο κ. Παστορούτη έχει το λόγο. Εντάξει, μπορείτε να ξεκινήσετε πάντως. Αλλά κύριο Παστορούτη, μπορεί να ξεκινήσει να μας κάνει την εισήγησή του ή μήπως χρειάζεστε εδώ το υλικό για τον υπολογιστή σας. Δυστυχώ δεν διαθέτουμε χρόνο. Σε 20 λεπτά θα πρέπει να κλείσει. Μη σα διακόψω λοιπόν. Α, η μοίρα, η μοίρα η μοίρα. Ε, θα, θα έρθει ο τεχνικό μεταξύ αυτό, μήπω μπορείτε ξεκινήσετε και θα σα έρθει βοηθώντα και ο τεχνικό. Ε, καλό απόγευμα, κυρίε και κύριοι και μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και τη Επιτροπή. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω γιατί μα δώσατε, μα προσφέρετε την ευκαιρία να σα πούμε για ποιου λόγου υποβάλαμε αυτή την αναφορά. Πριν να μπούμε τώρα να επιστρέψουμε σε λεπτομέρειε του θέματο, να τονίσω κάτι δεν μας προσκάλεσαν επίσημα στη σημερινή συζήτηση της ε, έκθεσης αναφοράς. Μόνο χθες ε, από τους φίλους της Βαλσούζα μας ενημέρωσαν ότι θα συζητιόταν σήμερα το δικό μας θέμα θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα. Δεν μας επέτρεψε να έχουμε και τα κατάλληλα στοιχεία τα οποία όμως στη συνέχεια θα σας αποστείλουμε. Η αναφορά μας έλεγε ότι αυτό το κομμάτι, το μέρος του διαδρόμου 5 θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί. Που είπαμε ότι πρόκειτο για τρέλα, καθαρή τρέλα, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσαμε. Τα γεγονότα απέδειξαν ότι είχαμε δίκιο. Ήδη σταμάτησε από την άνοιξη του 2010 η πραγματοποίηση ενός κομματιού και στην Τεργέστη, Η Τεργέστη εξαφανίστηκε από τη σημερινή χάραξη εάν μας είχαν ακούσει στην Ευρώπη τότε έγκαιρα, τότε δεν θα χανόταν ευρωπαϊκό κονδύλια που πήγαιναν για ένα σχέδιο που πήγε μετά στο καλαχτώνα χρήστων. Και δεν γνωρίζουμε ούτε ποιο ήταν αυτό το ποσό. Και ο αρμόδιος, ο διοικητικός Ρικάρντο Ρικάρντι, δημόσια αρκετές φορές το υπερασπίστηκε πολιτικά, διοικητικά, θεσμικά. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να προσέξουμε τη σημερινή ανάλυση που έχει να κάνει με το κομμάτι ε, Βενετία τεριέ τη υψηλή ταχύτητα και με το κομμάτι μετά τα σύνορα τεριέ τη Διβάσα αντικείμενο τη αναφορά μα στην περιοχή του Βένετο. Αρκετοί δήμαρχοι είπαν ότι θα πρέπει να πάει προς το εσωτερικό αυτή η γραμμή, η οποία δεν έχει χαραχθεί ακόμα δεν έχει σχεδιαστεί. Και αυτό για να μην πάει παράλληλα με τον, ε, διεθνή, τον εθνικό δρόμο, για το Στράντα. Εδώ με μια ευθεία 20-30 μόνο χιλιόμετρων δεν μπορεί να είναι αυτή η γραμμή ε, υψηλής ταχύτητας στο μέρος Πορτογκουάρο Ρόνκι Ντελετζονάρι δεν ε, συμφώνησαν οι Δήμη. Και επίσης εδώ και εκεί κόβονται κομμάτια, δείγματα, έτσι καταχρηστικά σε αυτές τις περιοχές, χωρίς άδειε, χωρίς εξοδοτήσεις και αυτό για το κλείσιμο του σχεδίου για να υποβληθεί στις 31 μέχρι 31 12 του 2010 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος το 2005 απέρριψε αυτό το κομμάτι Ρον Πορτογκουράρο Ρονκί Γιατί προβλεπόταν αρκετά χιλιόμετρα σύραγγες απορρίφθηκε, υπήρχαν προβλήματα και δυσκολίες αξεπέραστες ε, και τρομερές προβλήματα ε, στους υδροφόρους ορίζοντες ε, στα ύδατα της περιοχής. Τρομερές επιπτώσεις στο περιβάλλον από αυτό το κομμάτι και λέει ότι το καρσικό σύστημα θα φυγόταν και θα άλλαζαν τα χαρακτηριστικά της περιοχής που είναι όπως ακριβώς και στο κομμάτι Τεργέστη διδάτσα. Και υπάρχει ιδιαίτερη παρουσία σπηλαίων παρατηρείται. Κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο περίπου δύο σπήλαια. Άρα λοιπόν η επεύθυνη ε, ο υπεύθυνο ε, μηχανικός Κάρλο Κόμιν ε, υποστήριξε αυτό ότι δεν υπάρχει ανάγκη παρομοίου δικτύου σε αυτήν την περιοχή γιατί ακόμα το κλασικό παραδοσιακό κομμάτι μπορεί να ενισχυθεί και να αρκέσει. Ίσως, ίσως, αλλά να περάσουν πολλά χρόνια ακόμα, ίσως απαιτηθεί αυτή η γραμμή. Και ακόμα ο Ρικάρντο Ρικάρντι από την περιοχή του Φριούλη χάραξε μια γραμμή, ένα σχέδιο για την έναξη του προγράμματος σε μερικά χρόνια και προβλέπονται ορισμένες δεκάδες χιλιόμετρα σύραγγας εδώ και εκεί με τρομερά υψηλό κόστος, εκατομμύρια ευρώ και ε, κοντά κοντά με τη σημερινή γραμμή που είναι επιφανειακή αυτή η γραμμή και από την οποία περνάνε δύο εμπορικά τρένα και μερικά επιβατικά τρένα μόνο την ημερησίως και αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχει υποδομή απαραίτητη, αλλά δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει πελάτης. Και ε, στο εμείς δεν χρειαζόμαστε νέες ε, γραμμές ε, υψής ταχύτητας, αλλά χρειαζόμαστε μία αναδιάταξη του συστήματος με νέο ε, υλικό, νέα τρένα, καλύτερες υπηρεσίες και επίσης συντήρηση του δικτύου για να αγγιθούμε και την ασφάλεια. Δεν θέλουμε χρήματα ευρωπαϊκά για αυτά τα συνδρομικά έργα που να προκαλέσουν τρομερά, τρομερές ζημιές στο ευαίσθητο και τρομερά όμορφο ταυτόχρονα αυτό οικοσύστημα. Και όλα αυτά που να επιβαρύνουν ε, δημοσιονομικά ε, και την Ιταλική πλευρά και να υπονομεύσουν και το δημοσιομικό πρόβλημα της Ευρώπης όπως συνέβη με την Ελλάδα. Και στον 884 το Ευρωκοινοβουλίο και Ευρωπαϊκής Επιτροπής απόφαση βρίσκομαι στοιχεία που μας ενισχύουν και αναφέρω συγκεκριμένα εφαρμόζοντας κριτήρια που να συμπεριλαμβάνουν ε, απόψεις περί απόδοσης οικονομικής ε, την και τη δυναμική τους. Ζητάω μια, ένα έλεγχο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διαφωτίσει τις πτυχές αυτές, το σκάνδαλο αυτό, να ακούσουν και τις περιφέρειες αλλά και τους ντόπιου δήμαρχους επειδή δεν υπήρξε διαφάνεια και ακόμα και τις επιτροπές που έχουν δραστηριοποιηθεί επί τόπου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κάτι θα θέλει να προσθέσει σίγουρα σε αυτά που είπε προηγουμένως. Μπάρκερ. Eh, Δεν έχω πολλά να προσθέσω στο όσα είπα πριν. Η Επιτροπή πήρε πολλές πληροφορίες σχετικά με την αναφορά αυτή από τον Απρίλιο του 2010 αλλά ήδη είχε ξεκινήσει από νωρίτερα, από το 2007. Γράψαμε την 1η Οκτωβρίου του 2007 στον αναφέροντα γιατί έστειλε αντίγραφο τη επιστολή σε διάφορους επιτρόπους, οπότε απαντήσαμε και στην επιτροπή σας. Σήμερα επιβεβαιώνουμε τη θέση που παρουσιάσαμε εδώ το 2008, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία απόδειξη παραβίασης τη νομοθεσία για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των πληροφοριών που μας έχουν φτάσει και υποβληθεί. Επίσης, δεν ε, υπάρχει τίποτα για το, από το Πορτοκάγιο μέχρι το Τιβάτσο που να έχουμε δεχτεί. Δηλαδή υπάρχουν τρία τμήματα για τα οποία δεν έχει δοθεί καμία ε, έγκριση για αναπτυξιακά σχέδια. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν. Άρα πρέπει να φτάσουμε πρώτα στην αναπτυξιακή πτυχή και μετά να αποφασίσουμε κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει παραβίαση της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές ε, επιπτώσεις. Είναι υποχρεωτική η ε, εκτίμηση αυτή επιπτώσεων για τα τρία τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια μελέτη και επειδή πρόκειται και για ένα διασυνοριακό τμήμα πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας αυτής και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που έχουν να κάνουν και με τη Σλοβανία και με την Ιταλία που είναι και οι δύο χώρες μέλη. Η οδηγία δεν απαιτεί μελέτη για το κόστος και τα κέρδη, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά. Πρόκειται για περιβαλλοντική οδηγία. Σχετικά με το Natura 2000, το Κάσο, στο Κράτος, το Βιλάριο, στο Λαγκούνς, πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση βάσει των διατάξεων της οδηγίας Habitat. Και θέλω να ολοκληρώσω με αυτά που έχουν πει και οι συνάδελφοι ότι κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση είτε στηρίζεται από τα θεωρητικά ταμεία είτε από τον προπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων πρέπει να ε, σέβονται την νομοθεσία για το περιβάλλον. Δεν έχουν πάει χρήματα για το τιβάτσα παρά μόνο για προκαταρτικές μελέτες. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, πάει με αποστολή επιτόπου εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση. Αυτό θα ξεπέρναγε τις αρμοδιότητες μας βάσει των συνθηκών. Θα τις υπερεύαινε και δεν θέλουμε. Grazie, Στο Κονελιάνο κατοικώ εγώ, κοντά κοντά, στην περιοχή αυτή, για την οποία συζητάμε τώρα. Και όταν μου δώσατε αυτό το φυλάδι όταν μπήκα στην αίθουσα, με ξέπληξε η άποψη των πολιτών. Δύσκολο να έχουμε αυτό τον τίτλο ορισμένων πολιτών γιατί και εγώ, μια και είμαι εκεί κοντά, είμαι μέρος της γενικής γνώμης των πολιτών. Αλλά λοιπόν όχι των πολιτών, μέρος των πολιτών. Αυτό για να πούμε πώς έχει το θέμα. Εμείς έχουμε αναλάβει υποχρέωση απέναντι στις εκλογές μας και αυτό που επιθυμούμε και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιτελέσουμε το έργο μας και μάλιστα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν τα σκεφτόμαστε τα πράγματα, ποτέ δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Δεν ξέρω μήπως χαρακτηρίζει αυτή η συμπεριφορά την Ιταλία ή κι άλλους εδώ και εκεί είναι διάσπαρτη αυτή η συμπεριφορά στην Ευρώπη. Μήπως είμαστε εμείς κάπως ε, ειδικοί, special στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Ορισμένοι δίνουν τη μάχη τους ε, η Ευρώπη να μας προσέξει και άλλοι λένε όχι μακριά η Ευρώπη δεν το χρειαζόμαστε, δεν σας χρειαζόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι παίζουμε εδώ μπρος πίσω, ένα βήμα μπρος, ένα πίσω. Πάντως είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι εντάξει για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια, όλα αυτά έτσι αλλιώς πρέπει να υπάρχουν. Ο ρόλος μου εδώ είναι διαφορετικό σε μένα. Αυτός ο διάδρομος PP6, ο πρώην πέντε διάδρομος να αποτελέσει πραγματικότητα. Μην το δούμε μόνο έτσι τοπικιστικά, εντελώ τοπικιστικά το θέμα. Από εδώ, από δίπλα, από πάνω, από κάτω και stop να μην μπορέσει να ανοιχτεί αυτός ο διάδρομος. Εγώ θέλω να το δω στο πλήρες σύνολο μέσα, μια ευρωπαϊκή διάσταση και στιγμή για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και μετά να προσπαθήσουμε να βρούμε και επιτόπου την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό το ταιριέ στην τιβάτσα αποτέλεσε καρπό συζητήσεων, συναντήσεων, προσπάθεια συντονισμού και να μπορέσει να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις ε, και για μια λύση αποδεκτή σίγουρα έχει ζητηθεί από για πάρα πολύ χρονικό, μακρύ χρονικό διάστημα και, από, και να γίνει δεκτό από πολλούς, γιατί από όλους αποκλείεται ποτέ. Πάντως ε, πραγματοποιείται, προχωράει το σχέδιο, το πρόγραμμα και με την παρουσίαση του σχεδίου στις διάφορες φάσεις ε, σίγουρα θα δείξουμε ότι οι προδιαγραφές κοινοτικές τηρούνται, γίνονται σεβαστές θα θέλαμε να πούμε ότι δεν γίνεται και ούτε και εγώ θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο τώρα μην τα συμβαστούμε αυτά. Τώρα για το λόγο κόστους κόστους-οφέλους, το Cross 5 του 2008 για το εταιρεία στην Τιβάτς ε, δείχτηκε αυτό, υπήρξε, συντάχθηκε μια έκθεση ε, που στην περιφέρεια του Φρίουλη στην ιστοσελίδα δημοσιεύθηκε αυτή και τώρα έχει οριμάσει ο χρόνος, ισχύουν ακόμα περισσότερο αυτά. Τώρα μπήκε στη μέση και η χάραξη στην περιοχή του Βένετο και στην περιοχή του Φριούλη λίγο πιο πάνω και για τη διαδρομή που ακολουθείτε. Εγώ δεν είδα ακόμα τη διαδρομή πάντως. Κάλεσα τον Επίτροπο Μπρίγχορστ στην Τεργέστη και με τη διοίκηση του Βένετο και πιο βόρεια του Φριούλη και μαζί με τον αρμόδιο οργανισμό να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, επαναλαμβάνω. Τώρα το να πάμε παράλληλα με την τάδε γραμμή, με τον τρίτο διάδρομο, το ένα το άλλο, δεν μπορεί έτσι να ασκηθεί κριτική κατάλληλη για κάτι που δεν το γνωρίζομαι άλλωστε. Γιατί κανονικά μέχρι το Δεκεμβρίου της χρονιάς αυτής του 2010 είχαμε πει ότι θα βασιόταν αυτά και ελπίζω πολύ πολύ σύντομα να δω ποια θα είναι η χάραξη αυτή, η διαδρομή αυτή. Αλλά η προσπάθειά μας είναι να πετύχουμε μια λύση που όσο γίνεται λιγότερο να θίξει το περιβάλλον, να κοστίσει τα λιγότερα χρήματα, να γίνει δεκτή όσο γίνεται περισσότερο από πλευράς περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν ένα σχέδιο που ε, η, ε, ε, η περιφέρεια εκεί να μπορέσει να εξετάσει, να αντιμετωπίσει όσο γίνεται καλύτερα και νομίζω καλόπιστα ότι εργάζονται καλά αλλά προς το παρόν ε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ούτε μελέτη αξιοπιστίας. Άρα λοιπόν το αντιδρά κανεί έτσι νομίζω ότι δεν είναι σωστό και λογικό να το δούμε πρώτα και μετά να δούμε. Ε, μέχρι τις 31 Δοδεκάτου για να δούμε και τις περιφέρειες στην απόψή τους, να δούμε πώς θα γίνει δεκτό κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλώ την Επιτροπή, την Πρόεδρο και όλους. Εάν δεν καταρθώσουμε να πετύχουμε κάτι και να έχουμε απαντήσεις που να είναι πιστευτές, ε, λογικές, λογικές και σαφείς ερωτήσεις. Απαιτείται, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο πραγματοποίησης αυτού του διαδρόμου Πέντε. Όπως είπα πριν, το λέω τώρα και για αυτή την περιοχή, γιατί γνωρίζω εκεί καλύτερα και περισσότερο την κατάσταση. Ε, συνάδελφος. Θα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για το εξής πρόβλημα. Θέλουμε να εκτιμήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, να μιλήσουμε για τις συνέπειές τους, ενώ ακόμα δεν έχουμε την ε, μελέτη για τις περιβαλλοντολογικές ε, επιπτώσεις. Γι' αυτό και ζητώ και στους αναφέροντες αλλά και στην Επιτροπή να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να υποθεί. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στη φύση, στο περιβάλλον και βεβαίως την ίδια ώρα πώς θα επηρεαστεί η ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων που ζουν ε, στην περιοχή αυτή και ίσως να ξαναδούμε τον σχεδιασμό εφόσον βεβαίως έχουμε τις ε, μελέτες αυτές για τις επιπτώσεις τις ε, περιβαλλοντολογικές. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να παρακολουθηθεί από εμάς με μεγάλη προσοχή. Δεν θα εγκαταλείψουμε το θέμα αυτό. Είμαστε ακόμα στη φάση σχεδιασμού από ό,τι κατάλαβα και επαναλαμβάνω απαιτείται διαφάνεια και βεβαίως η αναλογικότητα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες υποχρεώσεις, τουλάχιστον εμείς εδώ σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να το εκτιμήσουμε με έναν τρόπο, τουλάχιστον εγώ το εκτιμώ με έναν τρόπο, και μπορούμε να εκφραστούμε κατά. Όσον αφορά ε, το πώς θα εκφραστούμε, χρειαζόμαστε κάποιες ε, πληροφορίες που δεν έχουμε ακόμα, ούτε καν για τη βάση του σχεδιασμού. Κάποιος άλλος που επιθυμεί το λόγο παρακαλώ, όχι. 30 δευτερόλεπτα εσείς να μας πείτε την απόψή σας. Πρόκληση, άντε, ένα λεπτό. Εγώ είπα 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, άντε να το κάνουμε ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν ξέρω, τρομερά εγωιστής θα ήμουν ε, να πω ότι είναι οι περισσότεροι οι πολίτες ε, που είναι κατά. Αλλά όχι, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Αλλά για ορισμένου λόγου από τις πτυχές αυτές ε, περνάει κοντά ή μακριά από το σπίτι μου. Αυτές οι σπατάλες αυτά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στην Ιταλία για την κατασκευή δικτύων υψηλής ταχύτητας τρένων ε, θα πρέπει να μας κάνουν να το σκεφτούμε αυτά. Το 2007 στο δημοσιονομικό κανονισμό βλέπουμε ότι αναφέρθηκαν 13 δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρωθεί το χρέος όλα αυτά τα χρόνια και τι είχαν κάνει, είχαν ανοιχθεί μόνο 200 χιλιόμετρα στην Ιταλία. Αυτή η γραμμή είχε ανοίξει μόνο για όλα αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν ε, μην ε, συνεχιστούν τα πράγματα τώρα και μετά εμείς από εκεί να διαπιστώσουμε τις περιβαλλοντικές καταστροφές στη Ρόνκη Τριέστε. Από τη στιγμή που είπαμε, διαπιστώσαμε ότι θα ήταν εις βάρος του περιβαλλοντολόγου της καρσικής ε, διαμόρφωσης του εδάφους εκεί και στο ίδιο στην Τεργέστη τη Διβάτσα και το ίδιο και τι θα γίνει με τις σύραγγες πώς θα ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Πριν από μερικά χρόνια, παρόλο που είχαν ε, γίνει μελέτες και από σπηλαιολόγους κλπ, ε, ανακαλύφθηκε το σπήλαιο ένα σπήλαιο που δεν περίμενε κανείς, ούτε δεν κανείς ότι θα υπήρχε σπήλαιο εκεί κάτω. Και κάτι ακόμα το τελευταίο, σύντομα σύντομα, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή ο κύριος είναι από την περιοχή του Βένετο, ο κύριος Ευρωβουλευτής, ε, εμείς ε, στις περιοχές δικές μας λέμε ότι η ανάλυση που κάνουμε είναι σαν να είμαστε πατέρας οικογένειας τώρα από τη στιγμή που έχουμε υπηρεσίες που δεν τα καταφέρνουν ε, γιατί να κατασκευάσουμε νέες γραμμές, γιατί να σπαταλήσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας. Από όσα άκουσα, νομίζω ότι το αίτημα αυτό έχει να κάνει με κάτι το υποθετικό μελλοντικό και σχετικά με μια ανησυχία που εκφράζεται για ένα σχέδιο που κανονικά όμως θα πρέπει να δούμε τις φάσεις πώς θα προχωρήσει την Επιτροπή λέει, που λέει ότι το κράτος δεν έλεγξε τι γίνεται ε, και δεν υπήρξε καμία παραβίαση. Τώρα έχουμε τη συνέχεια, τώρα τα κοιτάζει η Επιτροπή. Προς το παρόν δεν μπορεί να εκφράσει μια άποψη γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία για να μελετηθεί το πράγμα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποια πρωτοβουλία, δεν έχω κάποιο στοιχείο στα χέρια μου, το μοναδικό πράγμα που το μπορούμε να κάνουμε στη φάση αυτή είναι από τη στιγμή που συμφωνούν και οι συνάδελφοι με αυτό που εγώ υποδεικνύω, είναι να αποσταλεί μια επιστολή στις ντόπιε αρχές, τοπικές αρχές, ώστε να εξεταστεί καλύτερα το θέμα και να μπορέσει να υπάρξει δημοκρατική συμμετοχή στις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί σχετικά. Λοιπόν, ένα βιενικό σημείο μας στις τοπικές αρχές οι οποίες συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Συμφωνείτε συνάδελφοι. Α, ναι, τότε το κλείνουμε το θέμα. Και βέβαια ο αναφέρον από τη στιγμή που θα έχουμε νέα συγκεκριμένα στοιχεία που θα μας οδηγούν σε μια ανάγκη εκτίμησης, τότε μπορεί να υποβάλει και πάλι την αναφορά του. Επόμενη, το 12. Εύελιν Σλέγγλ, Αυστριακής Ιθαγένειας, εξ ονόματος της ε, πρωτοβουλίας Βίπταλ Λέμπενσβέρτες, σχετικά με την αντίθεσή τους προς τη βασική σύραγγα Μπρένερο, στον Μπρένερο. Ο κ. Λότε Γκάμπερ ε, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δαπανίσει χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων με τρόπο ο οποίος πλήττει. Όλοι ξέρουν ότι πρόκειται για μια διαδρομή η οποία ακολουθεί την διαδρομή που ακολουθεί ο αυτοκινητόδρομος που πάει από το Μόναχο προς τον Νότο εδώ και 20 χρόνια και με υψηλή ταχύτητα πλήττεται το περιβάλλον της περιοχής αυτής και την ίδια ώρα και για την Αυστρία και για την Ιταλία το οικονομικό βάρος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την σύραγγα Μπρένερ μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας, καλείται να αναλογιστεί η αυστριακή κυβέρνηση, το αυστριακό κράτος, με 24 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το άρθρο 171 όσον αφορά την εργασία και τη διαδικασία εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουμε ότι δεν έχει τηρηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν τήρησε τη διαδικασία. Είπε ότι έλεγξε με την τέταρτη έκθεση του πρώην Ευρωπαίου Συντοριστή Κάρεν Βαλμίρτ την βιωσιμότητα από οικονομικής απόψεως αυτού του έργου. Ο Κάρελ Βαλμίρτ αναφέρεται στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη λέγοντας ότι όλοι θα πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους και ότι τα ενεχτά ερωτήματα, τα ερωτήματα που ακόμη εκκρεμούν θα πρέπει να διαλευκανθούν. Το Ιταλικό Εντελικό Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από τρία χρόνια ανέφερε ότι η Ιταλική πλευρά δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το τμήμα αυτό που της αναλογεί. Η αυστριακή πλευρά ακόμη εκτιμά την σύραγα. Ο νέος συντονιστής, ευρωπαίος συντονιστής, Κόξ, έχει αναφερθεί στο ποσό του ενός δισεκατομμυριού, το οποίο βρίσκεται στο αποθεματικό για ε, την σύραγα, ότι το ποσό αυτό θα δοθεί ενώ ακόμα το σχέδιο δεν έχει προχωρήσει. Πρέπει να σας πω ότι στην Αυστρία δεν υπάρχει ούτε ένας ε, Αυστριακός πολίτης ο οποίος να στηρίζει αυτή τη στιγμή το ε, διάνοιγμα αυτής της σύραγγας. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους προγράμματα, ηλεκτροδότησης και ακόμα εκκρεμούν μελέτες. Το ερώτημα λοιπόν που θα ήθελα εδώ να θέσω είναι για ποιο λόγο τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δαπονηθούν για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απελευθερώσει αυτό το ποσό που βρίσκεται στο αποθεματικό, ενώ τόσο πολλά ερωτηματικά παραμένουν ανοιχτά. Και όχι μόνο όσον αφορά το οικονομικό τμήμα, το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί με σοβαρότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, καθηγητές, οι οποίοι θεωρούν ότι το κόστος αυτού του ε, προγράμματος, αυτού του σχεδίου, ξεπερνά τα πλεονεκτήματα εάν υλοποιηθεί. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία δεν είναι αποδεκτή. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να δαπονηθούν για κινητικότητα με μεγαλύτερο αποτέλεσμα, για την παιδεία και την κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση. Η μελέτη κόστους ωφέλους θα πρέπει λοιπόν να διεκπαιρεωθεί και η σημερινή ο σημερινός σχεδιασμός ε, για την σύραγγα αυτή όσον αφορά την υπάρχουσα σύνθεση μπορεί να αναβαθμιστεί με ένα ποσό το οποίο σήμερα υπολογίζεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα βλέπουμε ότι οι σιδηροδρομικές αυτές συνδέσεις υπάρχουν, είναι υπερφορτωμένες και ότι πρέπει να δημιουργηθούν καινούριε. Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων βεβαίως θα πρέπει να συμπληρωθεί με πιο σύγχρονες επενδύσεις. Τα προγράμματα υπάρχουν. Η σιδηροδρομική αναβάθμιση των ε, υπαρχουσών διαδρομών σε αυτός και θα είναι πολύ πιο οικονομική και αποτελεσματική. Επίσης θα πρέπει να γίνει και μια μελέτη περιβαλλοντολογική. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο διάλογος με τους πολίτες μπορεί να οδηγήσει σε μια αναδιάρθρωση και αναμόρφωση των ε, διευρωπαϊκών προγραμμάτων και των ε, δικτύων μεταφοράς, τα οποία βεβαίως και χρήζουν εξυγχρονισμού. Σήμερα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις υποχρεώσεις της που είναι η στρατηγική εκτίμηση και επαλήθευση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Επίσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και να μπορεί να τηρηθεί. Σήμερα βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός για το 2017 μας οδηγεί σε μεγάλα ερωτηματικά. Σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο της Ιταλίας βλέπουμε ότι σε 20 χρόνια ενδεχομένως μπορεί να έχει τελειοποιηθεί το έργο αυτό και το οποίο δεν θα είναι πλέον απαραίτητο και δεν θα είναι έργο προτεραιότητας. Σήμερα λοιπόν μπορεί η σύραγγα του Μπρένερ να ξεκινήσει με ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να το χρηματοδοτήσει. Έχει το δικαίωμα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να ελέγξει τον προορισμό και την βιωσιμότητα ενός έργου, να δαπανίσει χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου και σύμφωνα με το άρθρο 171 πιστεύουμε θα πρέπει να εκτιμήσει ορθότερα και βάσει πιο εμπεριστατωμένων μελετών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την βιωσιμότητα αυτού του έργου και το κατά πόσο μπορούν να τηρηθούν οι μελέτες και τα χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν τα σφάλματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν και να γίνει μια πραγματική μελέτη κόστος-οφέλιος. Οι πολίτες της Ευρώπης και οι φορολογούμενοι της Ευρώπης θα σας είναι ευγνώμονες ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει το λόγο. Thank you, President. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω την υπόθεση αυτή. Είναι μια υπόθεση που δεκάδες τώρα την συζητάμε. Δύο εκατομμύρια περνάνε από τον Μπρένερ κάθε χρόνο φορτηγά και ο κόσμος στην περιοχή θέλει να αλλάξει αυτό και να χρησιμοποιείται περισσότερο το τρένο παρά η σειρά αυτή. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο πάντως και το Κοινοβούλιο το σχέδιο ήδη το 1994 και το 1996 και μετά επιβεβαιώθηκε το 2004 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα μετά από τόσα πολλά χρόνια και έξι χρόνια μετά από την τελευταία απόφαση του 2004, το σχέδιο υπάρχει και μπορεί να υλοποιηθεί. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, περάσαμε από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήταν μια διαδικασία που κράτησε χρόνο, με διαβουλεύσεις, με βελτοποίηση του σχεδίου. Το ξέρετε από τις απαντήσεις της Επιτροπής. Και εγώ συμμετείχα σε ακροάσεις σε συναντήσεις με τους συντονιστές, με τους δημάρχους, με εκπροσώπους τους, ε, των τοπικών παραγόντων και θέλουμε τη διαβούλευση αυτή με όλους τους πολίτες για κάθε σχέδιο. Και εκεί που μένω εγώ έχουμε περισσότερα τρένα τώρα. Ξέρω τι σημαίνει μια τέτοια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πόσο πολύ τη θέλουν οι πολίτες. Έχω πει την ε, αναφέρουσα ότι είναι, δεν είναι θέμα χρημάτων. Το θέμα δεν είναι η υποχρέωση να έχουμε μια τέτοια μελέτη κόστους ε, και επιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν βασιζόμαστε σε παλιά σχέδια. Η Γερμανία, για παράδειγμα, κάνει μια νέα ανάλυση κόστους ε, και ωφέλους. Άρα λοιπόν γίνονται. Το ζητάνε και τα ελεγκτικά συνέδρια, και το ευρωπαϊκό και τα εθνικά. Δεν έχω λοιπόν να προσθέσω τίποτα άλλο. Το σχέδιο αυτό είναι έτοιμο να ξεκινήσει και ελπίζουμε ότι θα προσφέρει και τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε και ότι θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις για τον τοπικό πληθυσμό, πράγμα το οποίο βέβαια που μέχρι τώρα αμφισβητεί πολύ αυτός από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αν θα μπορούσε να συμπληρώσει κάτι ο συνάδελφος. Ναι, για την μελέτη αυτή η περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οδηγία αυτή δεν είναι αλήθεια, δεν εφαρμόζεται στις κατευθυντηρίες γραμμές των διευρωπαϊκών δικτύων. Πρόκειται για τα κράτη-μέλη, όχι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ντόρφαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν μιλώ σαν μέλος μόνο αναπληρωματικό αυτό τη Επιτροπή, αλλά και σαν πολίτη που μένει λίγε εκατοντόδε μέτρα από τη γραμμή του Μπρένερο και ακούει να περνάνε 220 τρένα ημερήσια και θα πάμε στα 400 τρένα όταν ανοίξει, συμπληρωθεί και το κομμάτι στην Αυστρία. Και είμαι και πρώην δήμαρχος ενός μιας πολιτιούλας στην περιοχή και που θα έχει και το μεγαλύτερο εργοτάξιο στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν ε, σαν αρμόδιος να υπενθυμίσω δύο-τρία πραγματάκια. Στο Μπρένερο άνοιξε στο 1865 μια αστυνομική γραμμή και επίσης η οτοστράτα του Μπρένερο το 1970, 100 χρόνια μετά, μέχρι το άνοιγμα της οτοστράτας, οι μεταφόρες γινόταν μόνο στο δρόμο στην στο, γινόταν πρώτα στην, ε, με το και μετά στο δρόμο. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί δεν επένδυσε κανείς ε, στους σιδηροδρόμους ε, αλλά μόνο στο δρόμο. Και τώρα σιδηρόδρομος παλιός 140 ετών με παλιά τρένα ηλικία 40-50 ετών θα πρέπει να ανταγωνιστεί ένα καινούριο διεθνή δρόμο με νέα φορτηγά κλπ και ο μοναδικός ε, τρόπος ε, για να ε, μεταφερθεί κανείς στη συνομική γραμμή θα πρέπει να κάνει το ίδιο όταν έγινε το αντίθετο, δηλαδή να πάει προς το να επενδύσει. Γιατί είπε η συνάδελφος προηγουμένως ότι και με την παλιά γραμμή ίσως θα μπορούσαμε να φτάσουμε τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Ίσως δεν είναι παρσάλπις τι γραμμές είναι κατασκευασμένες και στις τροφές τι δικές μας αν θέλετε να πάτε με 250 χιλιόμετρα την ώρα δικό σας το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται εκεί πάνω στα βουνά μας. να υπενθυμίσω δύο-τρία πράγματα γιατί αυτά που υπόθηκαν σήμερα σηκώνουν και ορισμένες διορθώσεις. Επαναλαμβάνω, τέλος πάντων, ε, τι διαβάζω στην αναφορά. Το τρένο έχει μεγάλη σημασία για τις μεταφορές στις Άλπεις. Το Μπρένερο, στο Μπρένερο και επιβάτες και εμπορεύματα αυξήθηκαν τρομερά. Τρομερά η κίνηση, το βάρος. Εμείς δεν το επιδιώξαμε, αλλά αυτό συμβαίνει παντού άλλωστε, στις Άλπεις. Αλλά φέτος μειώθηκε η μεταφορά παντού. Γιατί? Γιατί είχαμε παντού οικονομική κρίση, λοιπόν έχει κόψει κίνηση από παντού. Είναι όμως κάτι το προσωρινό, στιγμιαίο. Τώρα φτάσαμε πάλι στα 50 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων που ετησίως περνάνε από τη σύραγγα του Μπρένερο. Και σήμερα υπόθηκε ότι χρήματα δεν υπάρχουν, εκτός από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψευδές. Η Ιταλία πήρε κάθε απαραίτητη απόφαση για την χρηματοδότηση του έργου και η Αυστρία το ίδιο κάνει και ο δρόμος του Μπρένερο δίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του έργου αυτό. Λοιπόν υπάρχουν κονδύλια και μετά στην αφορά λέει ότι ε, δεν έχουν γίνει αναγνωστικές εργασίες. Μόνο για δύο μήνες όμως γίνει αυτό. Για γεωλογικά προβλήματα συχνά συμβαίνει σε παρόμοια έργα. Και ε, από την Ιταλική πλευρά δεν ξέρω. Από, απ' την ε, Ιταλική πλευρά έχουν προχωρήσει αυτές οι έρευνες και πριν από το χειμώνα θα έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και από την Αστριακή πλευρά που δεν ξέρω και τόσο καλά νομίζω ότι θα προχωρήσουν. Συνάδελφε, α, μισό λεπτό και ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Για το περιβάλλον. Ο πληθυσμός θα πρέπει να προστατευτεί από τα 400 τρένα τη μέρα. Άρα λοιπόν, η μοναδική λύση είναι να πάνε στη σύραγγα αυτά τα τρένα. Και επίσης θα πρέπει να προστατευτεί ο πληθυσμός από την εκπομπή ε, καυσαερίων από φορτηγά που 40 ας πούμε εκατομμύρια τόνοι εμπορεύματα, τα 10 πάνε στα τρένα θα πρέπει να προστατευτούν και εξοικονόμηση ενέργειας. Και με το καινούργιο θα αποφεύγουμε 700 μέτρα διαφορά επίπεδου. Είπατε ότι στην Αυστρία δεν υπάρχουν υπέρμαχοι από αυστριακής πλευράς για τον Μπρένερ και από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αντίπαλοι από ό,τι ξέρω τουλάχιστον και βεβαίως βασίζομαι πάντα σε σημειώσεις και άρθρα της ομάδας πρωτοβουλίας για την βιωσιμότητα της σύραγγας του Μπρένερ. Και από ό,τι ξέρω πολύ λίγα άτομα παραμένουν ακόμα αντίπαλοι. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε, αλλά πιστεύω ότι για κάποια θα πρέπει να εκφράσω τις αμφιβολίες μου. Παρακαλώ, σύντομα, σύντομα, γιατί ακόμα πλέον συνάδελφο Χέσλερ θα γίνει μια παρέμβαση και μετά να κλείσουμε. Αλλά απ' έξω μας περιμένει εδώ και 10 λεπτά ο Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής. Αλλά λοιπόν γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο όχι σαν τον προηγούμενο μιλητή. Δεν είμαι αντίπαλος ούτε των σιδηροδρόμων, ούτε της σύραγγας. Είναι πολύ λογικό αυτό, αλλά θα πρέπει να εξετάζουμε το κάθε σχέδιο συγκεκριμένα και είναι πολύ σωστή η ερώτηση του αναφέροντος αν είναι ορθό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δαπανά χρήματα φορολογούμενων στην Ευρώπη χωρίς προηγουμένως να έχουν εξεταστεί οι βλαβερές συνέπειες αυτού του έργου. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήματα και υπέρ και κατά. Εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να απαντηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα από την Επιτροπή. Στις 22 Απριλίου η απάντηση της Επιτροπής δεν είναι πλήρης και ούτε τώρα είναι πλήρης. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει μελέτη οικονομική κόστος ωφέλειας που βασίζεται σε σύγχρονα σημερινά στοιχεία και η οποία να δικαιολογεί ότι η χρησιμοποίηση αυτών των χρημάτων, των επενδεδημένων σε ένα τέτοιο έργο, θα αποφέρει ικανά αποτελέσματα και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια τέτοια μελέτη γιατί βάσει αυτής μπορούμε να αποφασίσουμε. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει σοβαρή πρόθεση χρηματοδότησης από μέρος των δύο πλευρών της γερμανικής των τριών μάλλον, της γερμανικής, της αυστριακής και της ιταλικής. Τρίτη ερώτηση. Η Επιτροπή έχει κάποιες προθέσεις όσον αφορά τα ποσά αυτά μέχρι το 2013 και τι προτίθεται να κάνει όσον αφορά την απελευθέρωση των ποσών αυτών που έχουν ε, σχεδιαστεί να επενδυθούν εάν, εάν επαναλαμβάνω, η προηγούμενη μελέτη δεν αποδείξει ότι είναι βιώσιμο το project. Μίλησα δύο λεπτά ενώ ο προηγούμενος ε, ομιλητής δέκα. Εγώ ζητούσα να δείξουμε κάποια ευγένεια και να υποδεχθούμε πως πρέπει τον ε, κύριο Διαμεσολαβητή. Παρακαλώ συνάδελφε, όσο γίνεται πιο σύντομα φτάσαμε σε αυτό και περιμένει και ο Διαμεσολαβητής ε, για να ασχοληθούμε το επόμενο σημείο. Ναι, ναι, θα σεβαστό αυτό που λέτε. Από αυστριακή απόψεω, πιστεύω ότι πρέπει να πούμε στην Επιτροπή ότι οι κοινότητε, στο Τυρόλο, το κρατήδιο, αλλά και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο Ντόρφμαν, το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού επιθυμεί να επιταχυνθεί αυτό το έργο και να φύγει το βάρος από τις σημερινούς τρόπους μεταφοράς. Καμία άλλη παρέμβαση. Δύο λεπτά. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον συναδελφό μου. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ωραία. Να σας πω το εξή. Επειδή ακούσαμε ερωτήσεις ε, για την Επιτροπή. Μήπως θα μπορούσε να μας απαντήσει γραπτός η Επιτροπή και μετά να δούμε στο τέλος ε, τι θα υιοθετηθεί σαν μέτρο για την ε, αναφορά αυτή στην οποία, για την οποία μίλησαμε γιατί δεν έχουμε χρόνο για να ακούσουμε άλλα και να απαντήσουμε αυτά. Εντάξει, συμφωνείτε, ευχαριστούμε, περιμένουμε τις γραπτές ε, απαντήσεις θα τις ανακοινώσουμε στη συνάντηση των συντονιστών. Και τώρα το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ε, ζητάω συγγνώμη από τον κύριο Διαμαντούρο για την ε, καθυστέρηση αυτή. Σχετικά με την πρόσβαση λοιπόν του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Νομολίου Συμβουλίου και της Επιτροπής, συντάκτρια τη, κυρία Χάνκης. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι περίπλοκο, γι' αυτό και θα μιλήσω στη γλώσσα μου, στα ουγγρικά, λέει η κυρία Χάνκης. Προηγουμένως βέβαια θέλω να ρωτήσω κάτι κυρία Πρόεδρε, πότε πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτηση αυτή, διότι δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ που να μην έχει χρόνο ο διαμεσολαβητής μας για να συζητήσει μαζί μας, έτσι κι αλλιώς τον κάναμε να μας περιμένει. Πριν ξεκινήσω λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Πέντε λεπτά έχω στη διάθεσή μου. Αλλά τότε δεν θα φτάσει ο χρόνος για να μιλήσει και ο κύριος Διαμαντούρος. Άντε 20 λεπτά. Γιατί μας έδωσαν, μας παραχώρησαν πέντε λεπτά η διερμηνή, αλλά λοιπόν έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Χάνκη. Θα είμαι σύντομη λοιπόν. Θα επικεντρωθώ στα κύρια ζητήματα. Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε τον ε, κοινό παρονομαστή μεταξύ διαφορετικών απόψεων και διαφορετικών πολιτικών ομάδων και όλοι να καταφέρουμε να συμβιβαστούμε και να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Αλλιώς θα βρεθούμε μπροστά σε μια μακρά διαδικασία, κάτι που δεν είναι ο στόχος μας. Θέλουμε μια καλή λύση. Ε, λοιπόν, υπάρχει ελπίδα για συμβιβασμό. Και αυτό γιατί εγώ πιστεύω ότι οι στόχοι και οι αξίες βάσει των οποίων θέλουμε να προχωρήσουμε και να δώσουμε πρόσβαση στην ε, πληροφορία για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι κάτι κοινό μεταξύ μας. Η στόχη είναι κοινή. Θα σας υπενθυμίσω μία πρόταση του κ. Διαμαντούρου που διάβασα σε κάποιο άρθρο όπου είπε ότι και σας το διαβάζω στα αγγλικά γιατί το άρθρο γράφτηκε στα αγγλικά, είπε το εξή λοιπόν. Αν οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή δίκηση είναι διάφανη, επιτυχής και λογοδοτή, τότε θα έχουν εμπιστοσύνη σε αυτή και θα θέλουν να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει η Ουγγρικά Ομιλήτρια, πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό. Η διαφάνεια η πρόσβαση και να ξέρουν τι να περιμένουν οι πολίτες. Αυτές λοιπόν είναι κοινέ αξίες, βάσει των οποίων πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που όπως είπα έχουμε μπροστά μας και να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβασμούς. Σύντομα λοιπόν τώρα, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ορισμένες πτυχές της γνωμοδότησής μου. Αρχικά η Επιτροπή το 2001 εκφράστηκε και στη συνέχεια και το 2008 και το 2009 τροποποιώντας το κείμενό της βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε πολλά μπροστά μας, πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Το πρώτο κριτήριο είναι η έννοια του τι σημαίνει έγγραφο, document. Και ε, λοιπόν, εδώ έχετε γραπτά όλη την τεκμηρίωση, οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις προτάσεις που γίνονται όσον αφορά τον ορισμό του τι είναι έγγραφο. Είναι σημαντικό πάντως ο ορισμός του όρου document, έγγραφο, να είναι επίσημο έγγραφο. Άρα λοιπόν το εύρος να επεκταθεί της έννοιας αυτής. Ποια έγγραφα δηλαδή είναι εκείνα στο οποίο έχει πρόσβαση ο κόσμος. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν πρέπει να φτάσουμε στα άκρα. Δεν θέλουμε να επεκταθεί η έννοια σε όλα τα έγγραφα που να είναι δηλαδή και σχέδια και μεμοράντα και τα λοιπά. Όχι, αυτά δεν λέω ότι πρέπει να είναι πράγματα στο οποία να έχει πρόσβαση το κοινό. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαραγωγικό, γιατί θα σήμαινε ότι συζητιούνται τα πάντα στους διαδρόμους, στα καφενεία και ότι τελικά δεν είναι γραπτά. Όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι η εξή. Όλα τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Άρα λοιπόν εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός και πρέπει να περιλάβουμε παντός είδους πληροφορίες βάσει του συστήματος αυτού. Το τρίτο σημαντικό ζήτημα για μένα είναι ο ορισμός του ε, συμφέροντος του κοινού. Εδώ υπάρχει η περίπτωση Μπαβάρια Λάγκε που γνωρίζουμε όλοι. Η Επιτροπή θα έπρεπε να επεξεργαστεί κατά τη γνώμη μου μια ομοιόμορφη θέση όπου να εξηγεί ποιο είναι το συμφέρον του κοινού. Λίγοι λένε ότι εδώ πρέπει να συμπεριλάβουμε τα πάντα και ότι όλα θα πρέπει να είναι ανοιχτά για το κοινό. Αλλά αλλού όταν πρόκειται για αντιτρομοκρατικές ενέργειες, SWIFT, PNR και άλλες συμφωνίες, είναι τέτοιες για τις οποίες εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προέχουν ε, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του ιδιωτικού βίου. Πρέπει να βρούμε δηλαδή μια καλή ισορροπία στην διατύπωση. Επίσης, το θέμα του απόρριτου να εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι δυνατόν το κάθε θεσμικό όργανο να αποφασίζει χωριστά τι είναι το απόρριτο και τι δεν είναι, τι είναι ευαίσθητο κλπ. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει πάνω σε ένα ενωπημένο σύστημα ορισμού των διαφόρων χαρακτηρισμών των εγγράφων. Έπειτα, η σχέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί. Τι είναι το τρίτο μέρος. Αν υποβάλει στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή έγγραφα, θα πρέπει να συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ρυθμίσεις. Έπειτα το θέμα του ανταγωνισμού και των σχετικών νόμων και αυτό πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο προβληματισμός της ενημέρωσης του κοινού επιδέχεται συζήτηση και οι παραβάσεις πρέπει να ακολουθούν την ομολογία. Έπειτα η μορφή πρόσβασης πρέπει να απλοποιηθεί. Πρέπει να είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να έχει πρόσβαση. Θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες εδώ για αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Λυπάμαι γι' αυτό. Πάντως έχω γενικά ε, διαφθρώσει την έκθεσή μου, αλλά αυτό το έκανα γιατί δεν είχα χρόνο. Ευχαριστώ. Eh. Διαθέτουμε ελάχιστο χρόνο και να μην διακόψω και στη μέση παρέμβασή του τον κύριο Διαμεσολαβητή. Γι' αυτό θα προτείνω να εργαστούμε μόνο στα αγγλικά. Άρα λοιπόν ε, να απελευθερώσουμε τους διερμήνες. Εντάξει και ο ίδιος ο κύριος Διαμεσολαβητής θα μιλήσει στα αγγλικά. Άρα λοιπόν να συμφωνείτε όλοι μας στα αγγλικά. Mr. Diamandouros. Madam Chair, thank you very much for making it possible for us to continue so that I will not feel that I'm taking the committee's time or your time.